Everybody who... Λοιπόν, όσοι δεν παρακολούθησαν την ε, συνεδρίαση ή δεν θέλουν να την παρακολουθήσουν μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα παρά το γεγονός ότι η συνεδρίαση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σας προτείνω να μείνετε. Ήσυχα όμως. So, I open now the Ξεκινά λοιπόν η συνεδρίαση της Επιτροπής Ίντα. Πρώτο σημείο της μερίσης διάταξης, η έγκριση. Ο κύριος Φίσας ζήτησε να αναβληθεί το σχέδιο έκθεσης το οποίο είναι για την επόμενη συνεδρίαση. Δεν έχω ε, κάτι άλλο να σας πω, γι' αυτό λοιπόν προτείνω να εγκριθεί η μερίσια διάταξη, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Σημείο 3, έγκριση των πρακτικών. Ως συνήθως, τα πρακτικά Τις της συνεδρίας 28-30 Αυγούστου θα εγκριθούν εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σημείο 4, παρομοίως, ανακοινώσει σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές της 29 Αυγούστου. Σημείο 5. Καταρχάς να σας πω πως ε, όντως ε, και αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Καλημέρα σας λοιπόν από το Λιούνεμπουργκ στο Ταλίν, στη Λισαβόνα, όπου μας βλέπετε από τις οθόνες σας. Έχουμε διερμηνία. Γι' αυτό σας παρακαλώ μιλήστε αργά, καθαρά και δυνατά για να μπορέσουν οι διερμηνείς να μεταφράσουν. Μετά, έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάντζεν, νέο μέλος της Επιτροπής, αντί... Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Την ξέρω, ξέρω τόσα χρόνια τη Βιβιάνε Ρέντινγκ και δεν μου έρχεται το όνομα. Έχει την ε, θέση της Βιβιάνε Ρέντινγκ από το Λουξεμβούργο. Και ο κύριος Χάνσεν είναι γεμάτος ενέργεια. Και ήρθε σε μας και στην αντιπροσωπεία της ε, Ιαπωνίας γεμάτος όρεξη για δουλειά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Καλώς ήρθατε. Μετά. περνάμε στην ηλεκτρονική μας ψηφοφορία. Η πρώτη έκθεση, την οποία θα ψηφίσουμε, η έκθεση για την τυθάσευση της παγκοσμιοποίησης και τις εμπορικές πτυχές αυτής. Ξεκινάμε ευθύ αμέσω μετά από δοκιμαστική ψηφοφορία, γι' αυτό λοιπόν ψηφίστε δοκιμαστικά. So we have still two members. Λοιπόν, δύο κάρτες. Λοιπόν, δύο μέλη που δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Test vote. Two members are not voting. So... Δύο μέλη δεν ψηφίζουν. Όπως και να έχει. Πέρας. Ξεκινάμε. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε την 42 ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Νομίζω εγκρίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 57. Πέρας. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβάστηκε 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 59 υπέρ, κατά απόχες απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές αυτό θέλει έλεγχο λυπάμαι κάθεστε τόσο μακριά σήμερα δεν σας βλέπω για να σας μετράω Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Είμαστε στην τροπολογία 66 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είχε εγκριθεί αλλά χρειάζεται έλεγχο αυτό. Ε, ηλεκτρονικά λοιπόν ψηφίζουμε την τροπολογία 69. And the vote is closed. Clearly adopted. Compromise 11. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 12 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, η 90 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 13α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 101 καταπίπτει. Η 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ως πιθανή προσθήκη είναι 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το επόμενα καταπίπτουν και πάμε στην 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τσεκ. Τώρα. Ελέγχουμε την 140 λοιπόν ηλεκτρονικά τώρα. Με αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ως προσθήκη 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Roll call. Ποιος ζήτησε ονομαστική κλίση. Ονομαστική κλίση στη συμβιβαστική 17α. 17 bis. Αρχίζει η ψηφοφορία. και Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Στο ελέγξουμε λοιπόν. 149 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Αλλά στο ξανά ελέγξουμε. 150. Αρχίζει η ψηφοφορία. και τελείων. Και εγκρίνεται. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Και εσείς τα ορεινά έδραν. 151. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά θέλει παρήθευση και αυτή. Ηλεκτρονικά λοιπόν επαληθεύουμε την 151. Αρχίζει ψηφοφορία και τελειώνει. Αγκρίνεται 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 153. Εγκρίθηκε σαφέστατα. Είχε 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Μάλλον έχει ζητηθεί ονομαστική κλίση για ένα τμήμα της τροπολογία αυτή και αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά Αποχέ. Ε, απορρίπτεται. Η συμβαστική 20 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά ας την ελέγξουμε καλύτερα. 183 αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και τελειώνει. Σαφέστατα εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Στην 190. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Mm, ισοψηφία. Αλλά απορρίπτεται. 191 είπε. Κατά. εποχές Έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε η ίδια ισοψηφία απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. 1919. Rejected. Ε, απορρίπτεται με την ίδια ισοψηφία. Κάτι λέξεις μικροφόνο η κυρία Κουίστατ. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε 39 μέλη παρόντα και ψηφίζουν τα 38. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγή δηλαδή. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος δεν ψηφίζει. Λοιπόν. Πού ήμασταν. Ε, συμβαστική 23. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 207 υπέρ κατά πίπτη. Oh my goodness. So, once again, two is seven. Πάμε πάλι, 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, 211 κατά αποχές απορρίπτεται. Η ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ τι θέλετε έλεγχο για ποια τροπολογία στην 23 Ωραία. η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα πέρας απορρίπτεται όπως σας είπα δεν με ακούτε συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές ορίστε Is there διαφωνεί κανείς να ψηφίσουμε όλες τις αιτιολογικές αναφορές μαζί. On block. Τα citations. Ναι, διαφωνεί. Ε, μία συνάδελφος, άρα όλα χωριστά. Η ένα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. δύο Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τρία Υπέρ. Κατά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 αποχές απορρίπτεται άκρη 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άκρη 12 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά πρέπει να το τσεκάρουμε ψηφίζουμε την τροπολογία 12 της Επιτροπής Γεωργίας αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση Πέρας. Νομίζω ότι είχε εγκριθεί όμως. Είδα πολλά πράσινα φωτάκια στα μηχανήματά σας. Επομένω συγκρίνεται. Και προχωρούμε. Άγκρι 16 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε τροπολογία 16 Επιτροπής Γεωργίας. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική πολίτευση. Πέρας. Τι θα γίνει με την περίπτωσή σας. <laughs> Απορρίπτεται. Ισοψηφία 19-19. Η άγκρη 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Άντε πάλι. Έλεγχος. Αρχίζει τώρα. Πέρασε. Α, απερίφθη τώρα σαφώς. Αγκρή 20 υπέρ. 100. Αποχές έλεγχος. 20 της Επιτροπής Γεωργίας. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Εγκρίνεται. Άκρη 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 26 υπέρ κατά αποχές Δεν σηκώνετε χέρια σας παρακαλώ υπέρ κατά Απόχες εγκρίνεται. 27 υπέρ. Πάντα της έγκρι. Ε, κατά. Απόχες απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται 34 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 35 υπέ, κατά απόχες απορρίπτεται 36 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 37 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 38 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. Καλτ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 11 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι είχε εγκριθεί. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 11 της Επιτροπής Πολιτισμού. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές και πάλι. Ε, σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Καλτ 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά στην την επαληθεύσουμε. Την τροπολογία 17 της Επιτροπής Πολιτισμού αρχίζει η ψηφοφορία και τελειώνει. Εγκρίνεται. Καλτ 19. Υπέρ. Κατά αποχές Ολόχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για τη 19 της Επιτροπής Πολιτισμού. Πέρασα. Εγκρίνεται. Η κάλτη 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάλτη 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά το ελέγξουμε καλύτερα αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η 30 της Επιτροπής Πολιτισμού ειπε Κατά. Αποχές. Και αυτό θέλει έλεγχο. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην ε, Επιτροπή Ανάπτυξης, τροπολογία 7, ΔΕΒ 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒ 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΤΕΒΕ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην 25 της Επιτροπής Αναρτική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η γνωμοδότηση Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Γιούρι 6, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι είχε απορριφθεί, αλλά στην έλεγξουμε καλύτερα. Εγκριθεί, λέει ο πρόεδρος τώρα, διορθώ. Εν πάση περιπτώσει, έλεγχος. Πέρας, εγκρίθηκε, ναι, Η Γιούρι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 9 υπέ κατά έλεγχος. The vote is open. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας απερίφθη. Γιούρι 10 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα το σύνολο του ψηφίσ... της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Okay. And the vote is... There is one too many. So one ε, περισσεύει ένας από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. And now the vote is closed. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία και κάτι αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. So. Λοιπόν, θα περιμένουμε για ένα λεπτό, έτσι ώστε όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα να μπορούν να το πράξουν, να κουβεντιάσουν και εσείς πίσω στη γαλαρία, έλατε πιο κοντά. So, dear colleagues in the back, please come a little bit closer. We have a lot of visitors today. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλατε λίγο πιο κοντά γιατί έχουμε πολλούς επισκέπτες σήμερα και πολλά σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Μετακινηθείτε λοιπόν, θα μας βοηθήσει. Okay, dear colleagues, so I reopen our... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινά ξανά η συνεδρίασή μας και περνάμε στο σημείο 5 της ανακοινώσεως του Προέδρου. Σήμερα είναι μία δυσάρεστη στιγμή στην ιστορία της Επιτροπής μας, διότι η Μύρια, η οποία εργάζεται στην Ίντα πάνω από 7 χρόνια, θα μας αφήσει. Φεύγει. Ε, είναι μία έμπειρη συνάδελφος, έχει καταφέρει να διεκπαιρεώσει πολλά σημαντικά θέματα και νομίζω πως θα μας λείψει πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε λοιπόν πολύ Μίριαμ για τη δουλειά που έχεις κάνει και καλή τύχη στη συνέχεια. Ευτυχώς δεν θα φύγει από το κοινοβούλιο. θα ε, πάει στην ε, Γραμματεία Συνδιαλλαγής και Συναπόφασης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν Μυρία Περνάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ σημαντικό νομίζω. Είναι η σχέση του εμπορίου και της τεχνολογίας blockchain. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτό το θέμα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που έχουμε αυτήν την ε, κοινοβουλευτική θητεία. Είναι και ένα από τα θέματα που έχει λάβει αρκετή δημοσιότητα εδώ και αρκετά χρόνια και νομίζω πως ε, έχει έρθει η ώρα να δώσω το λόγο στην συγχύτρια κύρια Μακλάρκιν για να μας πει περισσότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που δείχνετε τόσο ενδιαφέρον κύριε Πρόεδρε. Έχω λοιπόν την ευκαιρία να παρουσιάσω την έκθεση πρωτοβουλίας για το blockchain, μια μακρόπνοη εμπορική στρατηγική και να σας αναφέρω ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα και ζητήματα που είχαμε στην έκθεση. Είναι λοιπόν ένας τομέας εξαιρετικά ενδιαφέρον, και καινοτομίες λαμβάνουν χώρα καθημερινά και πιστεύω πως είναι ουσιώδε τα μέλη μας εδώ να ενημερώνονται όλο και περισσότερο. Ο κόσμος ε, μαθαίνει το blockchain και η τεχνολογία χρησιμεύει πέρα από τα bitcoin. Η έκθεσή μου λοιπόν θα εξετάσει το ρόλο και την αποστολή των blockchain στο διεθνές εμπόριο. σε σχέση με τα blockchain άδειε. Ε, ακριβώς ε, γιατί η τεχνολογία blockchain είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση του ότι καθώς αναπτύσσεται η τεχνολογία ε, θα εξελίσσεται η κατάσταση, θα μαθαίνουμε και περισσότερα. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα blockchain ιδιωτικών αδειών στο διεθνές εμπόριο και τους λόγους ε, για τους οποίους επέλεξα να εστιάσω αυτά τα θέματα θα τους βρείτε στο αιτιολογικό σημείωμα. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι εφαρμογέ του blockchain στο διεθνέ εμπόριο. Αναφέρομαι σε διάφορου τομεί όπου το blockchain μπορεί να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να βοηθήσει τι επιχειρήσει να αναπτυχθούν. Η έκθεσή μου λοιπόν εξετάζει πώ οι εμπορικέ πολιτικέ μπορούν να ενισχυθούν με την ενσωμάτωση του blockchain στη λειτουργία του. Για παράδειγμα, πολλέ φορέ ε, γίνεται λόγος για την ε, χρήση τους στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ε, στους κανόνες και προτιμησιακής πρόσβασης. Η διαδικασία λοιπόν χρήσης του blockchain θα βελτιώσει τη συμμόρφωση και θα κάνει τα ζωή μας πιο εύκολη. Γι' αυτό ως αποτέλεσμα θα τονώσει τις εξαγωγές μας. Θα ε, βοηθήσει επίση και στην, εμπορική, και στην αμυντική εμπορική πολιτική ε, με την ροή των αγαθών στην ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το, η εμπορική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναπτυχθεί με τη χρήση των διαφόρων πρωτοκόλων. Επίσης, η τεχνολογία blockchain θα εξυγχρονίσει τις δασμολογικές ποσοστώσεις καθώς θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στι τελωνιακέ αρχές και στους τελικούς πελάτες, έτσι ώστε οι ποσοστώσει να φαίνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και να υπάρχει περισσότερη ε, και καλύτερη πληροφόρηση για τα προϊόντα και για τις ποσοστώσεις. Επίσης, ε, το blockchain θα βοηθήσει στην ε, αύξηση της διαφάνειας, στην ενίσχυση της ε, παροχής και διάθεσης των αγαθών, στην αύξηση της προστασίας και της σταθερότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain, το διεθνές εμπόριο ε, μπορεί να αυξηθεί κατά 15%. Και επίσης, οι τελωνιακές αρχές θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν αυτόματα πληροφορίες ε, από πρωτογενείς πηγές για την ε, διακίνηση των αγαθών. Επίσης, η τεχνολογία blockchain θα μας απαλλάξει από την ανάγκη επιβεβαίωσης των στοιχείων και στα συστήματα ελέγχου των εισαγωγών αλλά και στα συστήματα των ε, επιχειρήσεων. Επίσης θα μειώσει τον ε, γραφειοκρατικό φόρτο και τον χρόνο που χρειάζεται για να ε, γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Επίσης, στην έκθεσή μου θα εξετάσω πώς το λογισμικό blockchain και τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας μπορούν να βοηθήσουν τα τελωνία και τις τελωνιακές αρχές να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα με την ε, μορφή της νομιμοποίησης εξώπεν από εγκληματικέ δραστηριότητες. Ε, επίσης, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε ε, και τα οποία ενδεχομένω εμποδίζουν τεχνολογία blockchain να ανθίσει. Αναφέρομαι στην ασφαλή ροή των δεδομένων, στα ε, παραποιημένα πλαστά έγγραφα και αγαθά που εισέρχονται στην αγορά και ε, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό γιατί είναι κέρια σημασία για το εμπόριο. Επίση, η τεχνολογία καταναμημένου καθολικού είναι πολύ σημαντική με συνδυασμό τη χρήση του blockchain και η έκθεσή μου αναγνωρίζει επίσης την ε, ανάγκη να εξετάσουμε το blockchain στο πλαίσιο του κανονισμού ε, προσωπικών ε, δεδομένων. Η τεχνολογία blockchain μπορεί να παρέχει λύσεις στην εφαρμογή του κανονισμού αυτού, ακριβώς διότι και, οι δύο, και τα δύο αυτά μέρη ε, διέπονται από τις ίδιες ε, αρχές. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στα προσωπικά και τα μη προσωπικά δεδομένα και να περιοριστούν οι επιπτώσεις ε, της ε, διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων στη χρήση τεχνολογίας blockchain. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει αυτός ο διαχωρισμός και επίσης υπάρχουν και δύο κύριες προκλήσεις στη χρήση των δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πρώτον, η διαλειτουργικότητα των διαφορών συστημάτων blockchain είναι πάρα πολύ σημαντική για να δημιουργηθεί ένα, αν θέλετε, οικοσύστημα με το οποίο θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε όλα τα ωφέλη του blockchain. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα γόνιμο περιβάλλον για τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, όπου θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία προς όφελός τους. Έπειτα, η πρόκληση που έχει να κάνει με την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain αφορά κυρίως την διεύρυνση των δικτύων ε, των εμπορικών δικτύων, ε, των τεχνολογικών δικτύων. Το σημαντικό είναι να δούμε ποιο πρωτόκολλο θα ε, επιλεγεί, γιατί, γιατί μπορεί μια χώρα να χρησιμοποιεί ένα και άλλη χώρα να χρησιμοποιεί άλλο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ομοιογένεια για να λειτουργεί η τεχνολογία blockchain με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, πρέπει να εξεταστούν οι πτυχές της εφαρμογής τεχνολογίας blockchain ε, και το πώς η τεχνολογία αυτή θα ε, βελτιώσει ε, την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των τελογινίων και θα αυξήσει τις εισαγωγές. Το blockchain μπορεί να αυξήσει την επικοινωνία και έχει τη δυναμική να διευκολύνει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Και τέλος, στις συστάσεις που κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες όπως ε, το παρατηρητήριο blockchain και τις διάφορες εταιρικέ σχέσει. Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις τη τεχνολογία και ε, επίσης τα πιλωτικά project που τρέχουν αυτή τη στιγμή σε διεθνέ επίπεδο, έτσι ώστε η βιομηχανία να ε, ενισχύσει την καινοτομία και να έχει διασφαλίσει ότι η τεχνολογία blockchain θα χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η συμμόρφωση και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να ε, έχουν ε, ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές, οι προκλήσεις και τα ωφέλη. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με την Επιτροπή, με εσάς εδώ, έτσι ώστε να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει σε ηγετική θέση καθώς ε, όλες ε, οι χώρες, όλο και περισσότερο, χρησιμοποιούν την τεχνολογία blockchain και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δράσει όχι μόνο στην ε, νομοθετική ρύθμιση, αλλά και στην ανάπτυξη και χρήση τεχνολογίας blockchain και ελπίζω η έκθεση αυτή να πυροδοτήσει συζητήσεις ανάμεσα στην Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Νομίζω πως ήδη το έχει κάνει αυτό και ελπίζω και προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψεων και ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς που ε, μετέφρασαν το τόσο τεχνικό κείμενο που είχα να σας παρουσιάσω σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακλάρκιν. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητές για δύο λεπτά, το πολύ στον καθένα σας. Κυρία Αντρική είναι για το ΕΛΚΑ, είναι πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαμακλάρκιν για την εξαιρετική της έκθεση η οποία πιστεύω αποτελεί άριστη αφετηρία για μας ε, για να διερευνήσουμε τις διάφορες δυνατότητες ε, για το πώς ε, τεχνολογίες καταναμημένου καθολικού όπως η blockchain μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της εμπορικής μας πολιτικής έρωτας τα εμπόδια και διευκολύνοντας τις εμπορικές διαδικασίες σε εποχές όπου το διεθνές εμπόριο βάλετε από παντού. Το blockchain αποτελεί μια φοβερή ευκαιρία για πιο διαφανές εμπόριο και πιο αποτελεσματικό εμπόριο όσον αφορά ε, το, τα, οικονομικά και για την άρση των εμποδίων. Για να έχουμε πιο ασφαλές και πιο αποτελεσματικό εμπόριο ε, χωρίς ε, τις έντυπες διαδικασίες που οδηγούσαν σε μεγάλες καθυστερήσεις σε όλη την αλυσίδα και πολύπλοκες διαδικασίες όπου ήταν ευάλωτε ε, σε απάτες. Οι λιανοπολιτέ, οι πολιτές χονδρικής ε, ε, θα μπορούν να γνωρίζουν καλά και να αξιολογούν καλά την ποιότητα των προϊόντων που πολλούν και αγοράζουν και θα υπάρχει και καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Αντικαθιστώντας τη γραφειοκρατία με τις τεχνολογίες αυτές, προβολή των πληροφόρων μέχρι το blockchain θα είναι αυξημένη και έτσι θα έχουμε καλύτερη προστασία των καταναλωτών, ενώ οι επιχειρήσει θα λειτουργούν καλύτερα με μητρώα και έγγραφα τα οποία δεν θα μπορεί να αλλάξει κανένα. Ιδιαίτερα τα μικρομεσαίε επιχειρήσει με την εισαγωγή του blockchain θα υποφεληθούν ιδιαίτερα και οι αναδυόμενε αγορέ επίση, επειδή ο χρόνο που δαπανάτε ε, στις εμπορικές διαδικασίες και στα έγγραφα θα μειωθεί και θα βελτιωθούν και θα απλοποιηθούν οι τελωνιακέ διαδικασίε. Το blockchain δεν είναι ε, το μαγικό ραβδάκι που θα μα λύσει τα πάντα αλλά θα βοηθήσει στο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στον σημερινό περίπλοκο παγκοσμιοποιημένο κόσμο παρέχοντα στου πολίτε και στου καταναλωτέ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή όμω παραμένουν ερωτήσει ε, ερωτηματικά και ε, κάποια πράγματα ασαφή. Χρειαζόμαστε περισσότερε απαντήσει να επιλύσουμε τα τεχνικά εμπόδια για την υλοποίηση των λύσεων blockchain. Πρέπει να έχουμε σωστή κανονιστική ρύθμιση και σωστού κανόνε προστασία δεδομένων. Επειδή πρόκειται για μια τεχνολογία σε εμβριακό στάδιο ακόμα, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, αλλά να μην προβούμε σε υπερβολικές ρυθμίσεις και παρεμποδίσουμε την πρόοδό τη. Επειδή υπάρχουν πολλέ δυνατότητε μέσα αυτή τη τεχνολογία για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρ Γκάμπελιτ, για του σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεση, το οποίο χαρακτηρίζεται από ισορροπία, θετική αντιμετώπιση γενικότερα επιδιώκει να φωτίσει περισσότερο την τεχνολογία blockchain και τις πιθανές της εφαρμογές στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Συμφωνώ με την κυρία Μακλάρκεν. Είναι ύψη τη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ε, στην πρώτη γραμμή και να προσαρμόσει την εμπορική της πολιτική στην ψηφιοποίηση. Αυτό είναι αναγκαίο για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασία σε έναν όλο ένα και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Η στιγμή λοιπόν είναι πρόσφορη να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς την Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας blockchain για ευκολότερη, αποτελεσματικότερη, ε, αποτελεσματικότερο ε, παγκόσμιο εμπόριο. Ωστόσο, να ξέρουμε ότι η τεχνολογία blockchain δεν αποτελεί πανάκια. Ο τομέας του διεθνούς εμπορίου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το blockchain σε διάφορους τομείς, ε, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει σε ποιου τομείς θα υπάρξουν ωφέλη και τι ωφέλη. Υπάρχουν κάποια πράγματα όμως που θα ήθελα να ενισχυθούν ε, στο σχέδιο έκθεσης. Πρώτα απ' όλα από πλευρά Κομισιόν ήθελα να τονίσουμε περισσότερο την ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης και έρευνας αυτό ώστε να αποκτήθουν περισσότερες γνώσεις και να διαδοθούν αυτές οι γνώσεις. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν κατευθυντήρες γραμμές ε, για την ε, ενδυνάμωση των εφαρμογών στους κατάλληλους τομείς που ε, μπορούν να υποφεληθούν πράγματι από αυτό συμβάλλοντα έτσι σε ένα πιο ασφαλέ περιβάλλον για τι επιχειρήσει που θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή σε εμπορικέ διαδικασίε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, διότι σήμερα έχουμε κανόνε και πρότυπα ε, που ενδεχομένω να είναι. Ε, ενδεχομένως σήμερα να είναι πολύ νωρί να εφαρμόσουμε κανόνε και πρότυπα. Ε, το κοινό, οι καταναλωτέ όλο και περισσότερο γνωρίζουν αυτέ τι τεχνολογίε, αλλά θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα που αγοράζουν έχουν παραχθεί ηθικά και βιώσιμα. Δεν πρέπει τα προϊόντα να παράγονται με κακέ εργασιακέ συνθήκε που βασίζονται σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ κλείνω επειδή μας σταματήσατε. Ευχαριστούμε πολύ η Νάντια Χίρς από το Άλντε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εισηγήτρια. έκθεση, το σχέδιο έκθεσης βγήκε πολύ καλό και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια γενική εικόνα ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο είναι το ελκυστικό σε αυτή τη τεχνολογία blockchain, ότι δεν μπορούν να τροποποιηθούν, να παραβιαστούν τα δεδομένα και δημιουργείται μια ε, αλυσίδα και για την διανομή και για την κυκλοφορία αρκετά ασφαλή και ε, στις εισαγωγές και τις εξαγωγές μπορεί να μειωθούν λοιπόν οι δαπάνες για την αποθήκευση των ε, δεδομένων και την εξασφάλιση τους. Ακριβώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μειώνεται το κόστος που είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Επίσης οι τελωνιακές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τις συναλλαγές και αυτό σημαίνει ακόμα ε, μικρότερο κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διεκπαιρέωση όλων αυτών των διαδικασιών. Εάν ε, χρησιμοποιηθεί και εφαρμοστεί καλά και σωστά αυτή η τεχνολογία είναι απόλυτο κέρδος. Αλλά χρειάζεται και ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο και είναι πολύ σημαντικό να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ιδιαίτερα με στόχευση το εμπόριο. Δεν βοηθάει να έχουμε τώρα εδώ αφηρημένες συζητήσεις, αλλά πάρα πολύ συγκεκριμένα να επικεντρωθούμε στο εμπόριο έτσι ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτή τη τεχνολογία. Εμείς έχουμε κάποιες μικρές ε, παρατηρήσεις ε, που θα κάνω και σχετικές τροπολογίες Θέλουμε να ενισχύσουμε το πεδίο εφαρμογή αλλά και τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μεγάλη πρόκληση. Βεβαίω και τα νομικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των δεδομένων. Θα κάνουμε κάποιες τροπολογίε, επαναλαμβάνω, αλλά σταματώ εδώ. Ε, ευχαριστώ ε, από τους Πρασίνους ο κύριος Μπίχνερ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ ε, την εισηγήτρια και δεν είναι τυπικέ ευχαριστίε. Αυτέ είναι ουσιαστικέ λέει ο κύριο Μπούχνερ. Η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή αφετηρία για μια συζήτηση σε βάθος. Πολλά είναι τα σημαντικά θέματα και τα πεδία εφαρμογής που ήδη αναφέρονται. Για μένα ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η διευκόλυνση του εμπορίου και η ελάφρυνση του εμπορίου, ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, η δυνατότητα καταπολέμησης ή περιορισμού καλύτερα και συστηματικά της ε, διαφθοράς και διαφόρων παρανομιών. Ε, ιδιαίτερα ε, αυτή η τεχνολογία blockchain. ε ιδιαιτερα αυτη η τεχνολογία αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε περιπλοκή των διαφόρων εμπορικών οδών. Σκεφτείτε κάποιες ψηφιοποιήσεις που δεν πήγαν καλά. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε ε, ορόσημα και ε, όπως είπε και η συγκήτρια, να φροντίσουμε να εφαρμόζεται σωστά η τεχνολογία. Αυτό ήταν το ένα. Ένα δεύτερο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η προστασία των δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πληγούν ε, αυτά τα είπε και η κυρία Μακλάρκιν. Παρόλα αυτά θα κάνω τροπολογίες ακριβώς σε αυτό το τομέα και χαίρομαι και προσβλέπω στην καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπεγκίν. Grazie Presidente. Colleghi, applicare la blockchain al commercio Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στο διεθνές εμπόριο είναι μια πρωτότυπη καινοτόμως ιδέα. και αυτό λοιπόν θέλω να δω την Ευρώπη μπροστά, πρωτοπόρο. Η τεχνολογία blockchain διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και καθιστά αδύνατη την ε, παραποίησή τους αν σκεφτείτε τον τρόπο που λειτουργεί ένα διεθνές σύστημα ανταλλαγή δεδομένων, μπορείτε να καταλάβετε πόσο μπορεί να βοηθήσει το blockchain. Και στα τελωνία και στον πόριο γενικότερα και για τις άδειε ε, στα τελωνία, έτσι ώστε οι τελωνιακές αρχές και ε, οι παραλήπτες των αγαθών να συνεργαστούν. Πέραν αυτό, σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και της ε, μεταφοράς ε, ενός προϊόντος, το σύστημα blockchain θα βοηθήσει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την προέλευση του προϊόντος, ώστε να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η παράνομη εισαγωγή. Όσον αφορά τις εξαγωγές, η blockchain θα μπορεί να βοηθήσει τους εξαγωγείς. Απλοποιεί τα έγγραφα, τα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία θα πάψουν να υπάρχουν. Θα μειωθεί έτσι το κόστος των εξαγωγών και θα αξιοποιούνται πλήρως οι εμπορικέ δυνατότητε που δεν γνωρίζουν συχνά οι επιχειρήσει. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την κυρία Μακλάρκεν. Είναι άριστη η έκθεση αυτή, αυτό το ψήφισμα και τη βλέπω πολύ θετικά. Και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες για βελτίωση του κειμένου και θα συμβάλλω και εγώ από το κίνημα των πέντε αστέρων σε αυτό το σημαντικό θέμα. Εύχομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να αναλύει πού θα είναι πιο πρόσφορη η εφαρμογή του blockchain στην εμπορική πολιτική και να μας, δώσει, να μας παρουσιάσει σύμφωνα ένα σχετικό έγγραφο. Οι δυνατότητες που προσφέρει το blockchain είναι αμέτρητες, δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Ξέρω ότι ποτέ η νομοθεσία δεν καλύπτει τα πάντα όσον αφορά τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά εδώ θα ήθελα να δω κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την Γκουε. κυρία Μινάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Έμα Μακλάρκιν και τους άλλους και ηγητές για τη δουλειά τους. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τεχνολογία αυτή η blockchain και ανοίγει ενδιαφέρουσε προοπτικέ. Αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που θα πρέπει να είμαστε πολύ επικριτικοί. Να σα αναφέρω ορισμένα πολύ σημαντικά για μένα. Οι bloggers έχουν το δικαίωμα και στη λύθη αυτό πώς ε, συνάδει με το blockchain, ότι βάζεις σε μια τέτοια λυσίδα, παραμένει εκεί και διατηρείται και είναι η βάση όχι για την ανωνυμία αλλά για την ψευδονυμία. Δηλαδή τα προσωπικά σου δεδομένα υπάρχουν και ταυτότητά σου απλώς με ψευδόνυμο. Ό,τι έχεις βάλει εκεί είναι δημόσια στο όνομά σου αν κάποιος συνδυάσει τα στοιχεία αυτά. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα της τεχνολογίας blockchain. Και κοιτάξτε, έχουμε και τον κανονισμό, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Χρειάζεται ρύθμιση εδώ της τεχνολογίας blockchain. Είναι περίπλοκη τεχνολογία αυτή, χρειάζεται κωδικούς και είναι και ε, ευαίσθητη για κάποιους κακοπροαίρετους εμπειρογνώμονες. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται έλεγχος όταν γίνεται ο λόγος για τη χρήση από τις δημόσιες αρχές, όπως λέει η έκθεση, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και από δημόσιο κανονισμό. Ας πούμε, η τραπεζική κρίση ε, προέκυψε μεταξύ άλλων και γιατί είχαμε ε, δώσει υπερβολική εμπιστοσύνη στον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών. Ε, καλή είναι η τεχνολογία, βεβαίως θα πρέπει να τη χαλιναγωγούμε και να τη ρεγουλάρουμε με τους δικούς μας ελέγχους και τα ενία ε, που θα βάλουμε και τις εγγύησεις. Και τέλος, υπάρχει και ένα στοιχείο περιβαλλοντικό. Ε, γιατί χρειάζεται τεράστια δύναμη, ε, χρειάζονται υπολογιστές πάρα πολύ ισχυροί, άρα καταβροχθίζει τεράστια ενέργεια. Τι θα γίνει, εντάξει, τα χρήματα που θα τα βρούμε. Δεν είναι μόνο τα bitcoin, υπάρχουν και άλλες εφαρμογές Καλή είναι η στόχη της Συμφωνίας των Παρισίων, αλλά τι κάνουμε ε, σε τέτοιες πρωτοβουλίες που θα πρέπει όλα αυτά να ενσωματωθούν στο σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσω το λόγο στον Λούκα Ντεκάρλι από τη Γενική Διεύθυνση Trade. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμμεριζόμαστε το ενδιαφέρον της Επιτροπής ε, για την τεχνολογία αυτή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως είπαν αρκετοί ευρωβουλευτές αυτό μπορεί να δώσει αρκετές ε, ευκαιρίες ε, και μπορεί να λειτουργήσει ως σημεία μια σφαίρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε, για, να δούμε όλες τις πτυχές της χρήσης του blockchain. Ένα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η τεχνολογία αυτή όταν εφαρμόζεται στο εμπόριο και στις αλυσίδες αξίας μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές όμως το blockchain δεν μπορεί να μας πει τίποτα για το πόσο αξιόπιστη είναι η πληροφορία ε, η οποία περιέχεται σε αυτό, την οποία κιόλας ε, εισάγουν οι χρήστες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε ποιος έχει πιστοποιήσει την πληροφορία και πώς. Ε, και με την αδειά σας κύριε Πρόεδρε θα ζητήσω από τη συνάδελφό μου Goodman να μας πει περισσότερα για την υποδομή του blockchain. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο. Και εμείς χαιρετίζουμε την έκθεση, η οποία μάλιστα ακολουθεί το σχέδιο που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2008 από το ε, FinTech. Μία από τις ε, πρώτες δράσεις που αναλάβαμε είναι να συστήσουμε ένα παρατηρητήριο το Φεβρουάριο φέτος ε, που ασχολείται με το blockchain με συμμετοχή πάνω από 1.500 ενδιαφερομένων από τον δημοτικό, ε, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εξετάζουμε περιπτώσεις χρήσης του blockchain και τις ε, αλυσίδες εφοδιασμού, που εκτός από τις άλλες εμπορικές πτυχές είναι μία, ένας, ακόμα τομέα, ένας ακόμα τομέας όπου χρησιμοποιείται πολύ η τεχνολογία αυτή. Επίσης, ε, εξετάζουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και σκοπός των εργασιών μας είναι να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς έχουν τα πράγματα, πώς εξελίσσεται η τεχνολογία και να ε, γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων ε, πρακτικών. Και ε, σε ό,τι αφορά την νομοθετική πλευρά για να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια δικαίου. Και Κάποια από τα σημεία που αναφέρατε ε, μας ενδιαφέρουν πολύ. Ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων ε, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε με μεγάλη προσοχή. Ε, γνωρίζουμε τις ανησυχίες που διατυπώσατε και ιδιαίτερα στην ομάδα εργασίας αυτή τη στιγμή ε, καταρτίζουμε μία έκθεση για το πόσο συμβατή είναι η τεχνολογία blockchain με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων. Θα τη δημοσιεύσουμε σε λίγες εβδομάδες περίπου. Κάτι άλλο που αναφέρατε και εδώ είναι η διαλειτουργικότητα οι πτυχές της διαλειτουργικότητας λοιπόν ε, εξετάζονται και στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης. Ε, συνεργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο για να εξετάσουμε ζητήματα διαλειτουργικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια. Έμα, ευχαριστώ πολύ όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τα σχόλιά τους. Πράγματι υπάρχουν προκλήσεις ε, και ευκαιρίες. Η τεχνολογία blockchain είναι περίπλοκη και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να την κατανοήσουμε και να την εναρμονίσουμε έτσι ώστε να άρουμε τους εμπορικούς φραγμούς, ε, να διευκολύνουμε το, εμπόλιο, το εμπόριο και τις ε, διεξαγωγές. Γι' αυτό λοιπόν για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος την τεχνολογία, το πώς χρησιμοποιείται όχι μόνο προς όφελος των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών για ένα εμπόριο το οποίο θα καταλαβαίνει, θα κατανοεί και θα χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνολογία. Και επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πρωτοπόρος να έχει ηγετική θέση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή της ε, χρήσης ε, της τεχνολογίας blockchain. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και να σας υπενθυμίσω ότι στις 11 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Γι' αυτό λοιπόν προσβλέπω στην καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι στις 11 Οκτωβρίου, μία το μεσημέρι, όχι 12, μία το μεσημέρι προθεσμία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και το επόμενο σημείο, το σημείο 8, αναβλήθηκε μέχρι την επόμενη ε, συνεδρίαση και περνάμε στο σημείο 9. αφορά την υπόθεση ενώπιον του ΠΟΕ για το Brexit και δίνω το λόγο στην κυρία Ρόβολ, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ξανασυζητήσει την έκθεση αυτή για την κατανομή των δοσμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ Έτη Ένωση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και τροποποίηση του κανονισμού αριθμό 32 κάθετο 2000 του Συμβουλίου. Ο τίτλο είναι αυτό τώρα τη έκθεση. Περί τίνος πρόκειται. Τα έχω ξαναπεί όλα αυτά. Ε, είναι μια πάρα πολύ τεχνική έκθεση. Και εξακολουθώ να θεωρώ κρίμα εάν αυτή η έκθεση αρχίζει να ισχύει μετά το Μάρτιο του 2019, όπου εμείς δεν θα έχουμε καμία επιρροή. Αφορά το ύψος των δασμών ε, που θα επιβάλλονται ανάμεσα στην Ευρώπη των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, βασική αρχή της μεθοδολογίας ποια είναι. Ε, θα πρέπει να τηρηθεί το σημερινό επίπεδο εισαγωγών-εξαγωγών έχοντας ταυτόχρονα όμως μια αντικειμενική βάση υπολογισμού όλων των συντελεστών των δασμών. Αυτό το θέλει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς ως ΕΛΚ δεν θέλουμε να πειράξουμε καθόλου αυτή τη μέθοδο. Το έχουμε πει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ τους συναδέλφους να μην αλλάξουν τίποτα. Ένας τεχνικός αργόριθμος είναι και ανάλογα με το προϊόν καθορίζεται ο συντελεστής ε, του δασμού. Τι, ποια είναι η πολιτική διάσταση εδώ πέρα. Πολλά μαθηματικά, λίγα πολιτικά. Για τα μαθηματικά δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Για τις τροπολογίε αυτό που είχε για μένα σημασία είναι ο αριθμός, ο, τρόπος υπολογισμού, η μέθοδος δηλαδή, να μην είναι ε, στις αιτιολογικές σκέψεις, στα recitals. Δεν έχει καμιά δουλειά εκεί. Αυτό είναι η ίδια η ουσία της έκθεσης. Θα πρέπει να μπει στα άρθρα. Ε, δεύτερον, πριν από μια επταετία περίπου, ο κανονισμός για την κατεξοδότηση πράξης τροποποιήθηκε ε, έγινε τεράστια δουλειά, θυμάστε με την οδηγία, οδηγίες όμνιμπους ε, και δεν συμμαζεύεται. Ε, αυτό όμως δεν φαίνεται στην έκθεση. Έχω κάνει αρκετές τροπολογίες λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση για να ε, ενημερωθεί, να επικαιροποιηθεί νομικά το κείμενο. Γιατί δεν κατάλαβα πάρα πολύ για ποιο λόγο το έτος 2018 ανατρέχουμε σε κάτι που ίσχυε πριν ε, την Omnibus ε, ως απόρρια της Λισαβόνας το 2010. Λοιπόν, οι δικές μου τροπολογίες δεν είναι τόσο πολιτικές, είναι μάλλον νομικής φύσεως ή τεχνικής φύσεως. Οπότε, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια νομοθεσία ε, γερή και αξιόπιστη. Ευχαριστώ πολύ, Γκοντελίβε. Σκιώδης ηγητές τώρα. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες απουσιάζει. Την Αλέσια Μόσκα την αντικαθιστά κανείς. Όχι. Η κυρία Μακλάρκιν από το ΙΣΙΑ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Είναι απαραίτητη μια καλή συνεννόηση ε, μεταξύ του Ηνωμένου Βασίλειου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσουμε του εμπορικού μα εταίρου ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στο εμπόριο με όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, να επεκταθεί λοιπόν το εμπορικό σύστημα όσο το δυνατόν περισσότερο. έχει αναλάβει ε, έχουν υποβληθεί προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα γίνει με τους δασμούς αφού αναχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, είναι μια ε, τεχνική άσκηση για την οποία οι διαδικασίες του ΠΟΕ παρέχουν τον απαραίτητο ε, μηχανισμό. Το ECR καλωσορίζει τι προσπάθειε τη εισηγητρία να διευκρινιστούν κάποιε από τι προτάσει τη Κομισιόν, όπω η μεθοδολογία που θα, στην οποία θα βασιστεί η κατανομή. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε, είναι σημαντικό να δείξει ευελιξία η Κομισιόν, ώστε η κατανομή να γίνει σωστά και να είναι υλοποιήσιμη. Επειδή ο μηχανισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί όμως σε περίπτωση απουσίας της συμφωνίας, μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα. Καλό την Κομισιόν να κάνει ό,τι μπορεί βάσει του άρθρου 28 του ΓΚΑΤ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρίτια δεν είναι εδώ. Κλάους Μπούχνερ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Όπως αναφέρθηκε ήδη είναι πολύ τεχνικό το θέμα αυτό και η συγγήτρια ακολουθεί τη γραμμή της Κομισιόν. Εμείς ως πράσινοι δεν έχουμε διαφορετική γραμμή και η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων, όσον αφορά την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων μετά από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρόταση θα κάνει την αλλαγή απλή σχετικά. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι πολλέ χώρε του ΠΟΕ θα έχουν να πούν τη δική του άποψη στη διαδικασία αυτή και δεν θα δεχθούν την πρόταση ε, κατανομής της Κομισιόν. Είχαμε μία πρώτη δήλωση ήδη από αυτή την άποψη. Εμείς ωστόσο ω πράσινοι συμφωνούμε φυσικά ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τέτοιου είδου ε, απόψει προ το παρόν εάν οι εταίροι του ΠΟΕ δεν έχουν πρόβλημα με όλο αυτό, θα πρέπει να αμφισβητήσουν, να υποβάλουν ένσταση ε, στη σχετικό μηχανισμό επίλυση διαφορών του ΠΟΕ. Οι περισσότερε τροπολογίε σε αυτό το σχέδιο έκθεση σχετίζονται με τη διαδικασία τη καταξιοδότησης και εκτελεστικών πράξεων για οποιαδήποτε αλλαγή στα προγράμματα ε, για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων ε, για τους εταίρους του ΠΟΕ. Εάν υπάρχει κάποια συμφωνία διαφορετική από την κλασική κατανομή. Η συγγήτρια Υπάρχει αντίφαση με την ποσόστοση του κανονισμού του 1992 και αυτό φαίνεται σε πρώτη ματιά ένας, μια μάχη νομική. Αλλά θα χρειαστούμε την απόκριση της Κομισιόν ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε κατά πόσο υπάρχει πολιτική ζημιά ως αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε τέτοιε συζητήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ από την ΚΟΕ, ο Χέλμοντ Σόλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ακόμα και αν ε, φαίνεται τεχνική έκθεση, έχει πάρα πολύ ευρείες ε, συνέπειες που φτάνουν μακριά. Γι' αυτό συμφωνούμε για τις της πράξεις. Δηλαδή το Κοινοβούλιο θα πρέπει πάντα να έχει λόγο και στις μελλοντικέ εξελίξεις των εμπορικών μας σχέσεων με τρίτες χώρες σε περίπτωση Brexit. Και ερχόμαστε αμέσως στην πολιτική διάσταση αυτής της τεχνικής ε, διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες επιπτώσεις του Brexit σε τρίτες χώρες εάν αυτό γίνει με τρόπο άτακτο και μη συντεταγμένο. και δεν καταλήξει σε μια αμοιβαία υποφελη συμφωνία η προσπάθεια αυτή. Είναι δύσκολο λοιπόν σήμερα να εκτιμήσουμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις και πού θα κινηθούμε. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Όλο αυτό το εγχείρημα λοιπόν είναι μάλλον μια προπαρασκευαστική νομοθεσία παρά μια οριστική νομοθεσία. Αυτό είναι το δικό μας σχόλιο από την ΚΟΕ για την αλλαγή του κανονισμού 32 κάθετος 2000 του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ματ Κάρθη ε, ε, είναι ο συνταξινομοδότης της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στην εισηγήτρια που με κάλεσε σε αυτή τη συνεδρίαση για να ακούσω τι απόψει τη επιτροπή και να μοιραστώ και τι δικέ μου μαζί σα. Πρέπει να πω ότι η Επιτροπή Άγκρη δεν έχει πραγματοποιήσει πλήρη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. Προτίθεται να το κάνει στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Θα σα μιλήσω λοιπόν ω εισηγητή τη δική μας γνωμοδότησης. Είναι σημαντικό το αρχείο αυτό για την Επιτροπή μα επειδή ο τομέα τη γεωργίας θα επηρεαστεί περισσότερο από όλου από αυτό το εγχείρημα επειδή κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων ε, αποτελείται ως επιτοπλίστων από γεωργικά θέματα, γεωργικά προϊόντα. Ε, έχει γίνει λοιπόν εκτενής αξιολόγηση του κατά πόσο οι ευρωπαϊκές αγορές θα μπορέσουν να απορροφήσουν αυτές τις δασμολογικές ποσοστώσεις ε, προς όφελος των προϊόντων που παραγόνται στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να πω ότι η επανακατανομή των ποσοστώσεων αυτών και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να αναγνωρίζουν πόσο ευάλωτα είναι ορισμένα τέτοια προϊόντα σε εξωτερικό ανταγωνισμό και φυσικά και τις ε, συνθήκες διαβίωσης των ε, παραγωγών. Αναγνωρίζω ότι η μεθοδολογία της Κομισιόν έχει συμφωνηθεί από κοινού με τους Βρετανούς εταίρους και ότι θέλει να ε, παρέχει τις παραχωρήσεις δίκαια για όλους τους εταίρους. Συμφωνώ λοιπόν με την εισηγήτρια. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να θεσμοθετηθεί στις διατάξεις ενός κανονισμού και όχι μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις. Από μόνη τη όμως δεν μπορεί να διασφαλίσει μελλοντική ισορροπημένη και δίκαιη κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων αφού όπω προειδοποιεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την εξουσία να αλλάξει αυτά τα νούμερα στο μέλλον. Όπως γνωρίζετε το Brexit ε, πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα και έτσι όπως ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις μπορεί να τροποποιηθεί ε, να τροποποιηθούν οι συμφωνίες για τις ασμολογικές ποσοστώσεις. Θεωρώ ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να έχει την απόλυτη διακριτική ευχαίρεια να αλλάζει την κατανομή χωρί ε, έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υιοθετεί ε, κατεξοδότηση πράξη μόνο εφόσον έχει συναυθεί πλήρω μια διεθνή συμφωνία. Για όλε τι άλλε τροπολογίε θα πρέπει να ε, υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει τη διαδικασία που θεσμοθετείται στι συνθήκε. Απουσία άλλη λύση και για να μην έχουμε τα σύνορα που φοβόμαστε στη Βόρεια Ιρλανδία, οι διαπραγματευτέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμφωνήσει ε, να παραμείνει η Βόρεια Ιρλανδία ε, στις, ε, στην εσωτερική αγορά και στην Τελωνιακή Ένωση. Αν γίνει αυτό θα πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις για επανακατανομή των TRQ όπως αναφέρεται στο παράρτημα και αυτό θα απαιτήσει πολιτικές αποφάσεις και θα πρέπει να περάσουν από κοινοβουλευτική εξέταση. Το μερίδιο των Βρετανικών TRQ είναι τόσο μικρό που η χρήση των ποσοστώσεων βάσει τη μεθοδολογία που προτείνεται θα δημιουργήσει παρόμοιε TRQ που μπορεί να θεωρήσουν οι εταίροι μας από το ΜΠΟΕ ανεπαρκές. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση και εκεί θα χρειαστούν πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να περάσουν από κοινοβουλευτική εξέταση. Σας δίνω απλά δύο παραδείγματα εδώ. Οπότε δημοκρατική εξέταση, κοινοβουλευτική έγκριση ή απέτηση διαπραγμάτευσης κάθε ε, συγκεκριμένης ε, δασμολογικής ποσόστοσης. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε κατανομή για κάθε κατανομή απαιτούνται όλα αυτά. Σκεφτείτε ποιε είναι οι συνέπειε των όσων μα ζητάει η Κομισιόν να εγκρίνουμε με αυτόν τον κανονισμό και με τι δυνατότητε τροποποίηση επανακατανομή στο μέλλον. Αναγνωρίζει έτσι πόσο σημαντικέ θα είναι οι συνέπειε κακών αποφάσεων ή αδιαμφισβήτητων ή μεροληπτικών αποφάσεων σε τέτοιου τομεί για του γεωργού ε, και τι τοπικέ κοινότητε σε ολόκληρη την Ευρώπη που θα επηρεάσουν το μέλλον των τοπικών οικονομιών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε από την Κομισιόν ο Μιχαέλ Νίαρ από την DJ Agri. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση, η οποία νομίζω μας δίνει μια ιδανική βάση για να οδηγηθούμε σε γρήγορη συμφωνία ανάμεσα σε όλα τα θεσμικά όργανα. Και με την άδειά σα ε, να αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα στο τέλο παρέμβασή μου. Συμφωνώ καταρχά με το ότι είναι πολυτεχνική πρόταση, τεχνική άσκηση, όμω έχει πολιτικό ενδιαφέρον και είναι πολύ λεπτό το ζήτημα πολιτικά. Αυτό φάνηκε και από την ομιλία του Πρόεδρου Γιούγκερ για την κατάσταση τη Ένωση νωρίτερα το Σεπτέμβριο, όπου αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα και ζήτησε μια γρήγορη συμφωνία. Διαβάζοντα την έκθεση, παρατηρώ ότι όλοι συμμεριζόμαστε τι ίδιε αρχέ και του ίδιου στόχου. Οι αλλαγέ λοιπόν τις οποίες προτείνει η συγγήτρια μου φαίνονται ε, αποδεκτές ε, και βέβαια ο τρόπο είναι το ζητούμενο. Όλοι έχουμε διαφορετικού τρόπου για να καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Νομίζω όμω πώ θα συνεργαστούμε επικοδομητικά και με εσά και με την Επιτροπή Γεωργία, έτσι ώστε να βρούμε μία λύση στα διάφορα θέματα που έχουν προκύψει. Τώρα, ε, πολύ σύντομα να αναφερθώ στα τρία σημαντικότερα για μένα σημεία. Πρώτον, μέθοδος. Όταν καταρτίζαμε την έκθεση, αναρωτηθήκαμε και εμείς το ίδιο. Η μέθοδος θα πρέπει να μπει στα άρθρα, στο διατακτικό και μετά να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την υλοποιήσει με συγκεκριμένα νούμερα ή να μπουν τα νούμερα κατευθείαν στην, ε, κυρίως, ε, στο, στο κυρίως ε, κείμενο, στο παράρτημα. Αποφασίσαμε το δεύτερο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τα νούμερα στο παράρτημα αυτή τη στιγμή και γι' αυτό έχει γίνει αναφορά στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις. Ακριβώς διότι μέσω του παραρτήματος έχουμε αυτά τα στοιχεία. Τώρα, αν θέλετε να μεταφερθεί η αναφορά αυτή στην ε, μέθοδο αλλού για την ανακατανομή των ποσοστώσεων, να μπει στα άρθρα δηλαδή από το παράρτημα, ε, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρέπει να το εξετάσουμε πρώτα και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση. Το σημαντικό είναι να γίνει μια σύνδεση της ε, μεθόδου με τα παραρτήματα, διότι από ό,τι βλέπω κανείς δεν θέλει να διαγραφεί το παράρτημα. Εκεί βρίσκονται όλα τα νούμερα, όλα τα στοιχεία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση έτσι ώστε όσοι διαβάζουν τον κανονισμό και πρέπει μετά να τον εφαρμόσουν να γνωρίζουν ακριβώς ποια δικαιώματα έχουν ε, σε τη φορά τις ε, εισαγωγές και το καθεστώς. Έπειτα, σε ό,τι αφορά την ε, ευθυγράμμιση του, 32, του κανονισμού του 32-2000 που ανέφεραν ορισμένοι από εσάς, Καταλαβαίνω και εκτιμώ το ότι 10 χρόνια μετά την θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχει έρθει η στιγμή να εναρμονιστούν οι βασικέ νομικέ πράξει που είναι πριν από αυτή. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι αυτή η εναρμόνιση δεν θα γίνει ούτε αυτόματα, ούτε είναι κάτι τεχνικό. Είναι μια πολιτική διαδικασία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πάντα την ίδια θέση ω προ τι λεπτομέρειε τη εναρμόνιση αυτή. Από ό,τι βλέπω, είπαμε για μία πλήρη εναρμόνιση του κανονισμού 32.000. Ε, Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που θα ήθελα είναι να κάνω μια παράκληση, να προσπαθήσουμε και με το Συμβούλιο να ε, συμβιβαστούμε, να περιορίσουμε κάπως εδώ την εναρμόνιση και να δούμε ποιο είναι το αναγκαίο για την πρόταση, το οποίο είναι να είμαστε αντικειμενικοί, να εργαστούμε αποτελεσματικά και να μην χρησιμοποιήσουμε την πρόταση αυτή για να γίνει συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές σε κάτι άλλο, και αυτό βασικό το οποίο όμως δεν συζητάμε σήμερα. Τρίτον, πεδίο εφαρμογή ε, των ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τροποποιεί τα παραρτήματα. εκτιμώ τις απόψεις σας ε, ε, και αναγνωρίζω το ότι εσείς θέλετε να μην έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν την αρμοδιότητα. Είστε, να είστε σίγουροι το Συμβούλιο το ίδιο σκέφτεται, οπότε νομίζω πως εκεί θα συμφωνήσετε. Ε, ένα μόνο να επισημάνω. Συμφωνούμε βέβαια όλοι για το ότι αν θέλουμε να συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας του ΠΟΕ στην Γενέβη για τη διαδικασία του άρθρου 28, Αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να ε, εκειωθούν από το Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο, από όλα τα θεσμικά όργανα και γι' αυτό νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να έχει την ε, δυνατότητα να τροποποιεί τα παραρτήματα. Ε, εκεί που ίσως είναι προβληματικό είναι στο σημείο Β, που αναφέρεται ότι θα λαμβάνονται υπόψη και άλλες πληροφορίες. Τώρα θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Δεν θέλουμε την εξουσία αυτή για να παρεκκλίνουμε από αυτήν την κοινή μέθοδο που έχουμε αναπτύξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Να είστε σίγουροι, σας διαβέω, δεν πρόκειται γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να το βάλουμε στο νομικό κείμενο θα το κάνουμε. Να είστε σίγουροι μαζί με τη δική σας συνεργασία και τη συνεργασία του Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, ε, στη Γενέβη, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μπορεί να προκύψει το εξή. Μπορεί μια τρίτη χώρα να μας ε, παράσχει αντικειμενικές ε, πληροφορίες, αλλά για πολιτικούς λόγους να μην μπορούμε να διηγηθούμε σε συμφωνία με αυτή την τρίτη χώρα. Μετά, αυτό που λέμε είναι ότι αυτές τις απτές πληροφορίες πρέπει να τις πάρουμε και να τροποποιήσουμε τα νούμερα στο παράρτημα έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για οποιασδήποτε νομικές διαφωνίες. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας, κοινό συμφέρον. Γι' αυτό και θέλαμε στο άρθρο 3 να συμπεριληφθεί και αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω, θέλουμε να συνεργαστούμε, όμως ε, σας κάνω έκκληση να μείνει αυτή η αρχή που μας δίνει ευελιξία, έτσι ώστε να ε, μπορούμε να, στο μέλλον να χρησιμοποιούμε καλύτερα τις πληροφορίες για να αποφεύγουμε νομικές ε, διαφορές. Τέλος, χρονοδιάγραμμα. Ξέρουμε όλοι πόσο επίγει το θέμα αυτό. Σας παρακαλώ να προσπαθήσετε με το Συμβούλιο να καταφέρετε να εγκριθεί ο κανονισμός πριν το τέλος του έτους θα έχουμε ελάχιστο χρόνο ακόμα στι αρχέ του 2019, όμω το χρειάζεται αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορέσει να εκδώσει τι ε, εκτελεστικέ πράξει για να γίνουν όλα αυτά πράξη. Γι' αυτό και το χρονοδιάγραμμά μα είναι πολύ ε, στενό. Πρέπει να κρυθεί μέχρι το τέλο του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Γκοντολίφ, έχει το λόγο. Είναι γεγονός φυσικά ότι είναι εν μέρη τεχνική αυτή η έκθεση, αλλά ό,τι έχει να κάνει με κατεξοδότηση πράξη ή εκτελεστικές πράξεις είναι ε, εξόχως πολιτικό και το ξέρουμε, δεν είναι τεχνικό θέμα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, λέω. Υπάρχουν αβεβαιότητες, το ξέρω, αλλά τη στιγμή της ψηφοφορίας δεν θα ξέρουμε ακόμα προς ποια κατεύθυνση ε, θα κινηθούμε ή με ποιο τρόπο θα γίνει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορούμε να το προσθέσουμε. Η προθεσμία δεν έχει λήξει ακόμα. Δεν έχει καν οριστεί. Βεβαίως είμαι διατεθειμένη και προφανέστατα να συνεργαστώ καλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο μετά από μια εμπειρία 30 ετών για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν θέλει να γράψουμε κάτι στην έκθεση... να μας ζητήσει επιταγή ελευκό να κάνει ό,τι θέλει το συντομότερο. Αλλά μετά τη Λισαβόνα εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε ενισχυμένη ε, ε, γνώμη να εκφράσουμε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, άρα και σε αυτό. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία και ελπίζω γρήγορα να φέρουμε σε αίσιο πέρα σε όλη αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν μπορώ παρά να το υπογραμμίσω και να το τονίσω αυτό, ότι από το 2009 και μετά έχουμε τελείως διαφορετική κατάσταση ως Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Μπορεί το θέμα αυτό να πιέζει πολύ χρονικά, αλλά εμεί δεν θα κάνουμε εκπτώσει τώρα στα δημοκρατικά δικαιώματα, ούτε θα τα θυσιάσουμε. Είναι σαφέστατο ότι θα προχωρήσουμε με βάση τις δυνατότητες ή διαμόρφωση των αποφάσεων που έχουμε. Προθεσμία για την καταθεση τροπολογιου τροπολογιών 5η Οκτωβρίου, 12 ακριβώς το μεσημέρι. Then we have uh, Τώρα έχουμε μια κοινή συζήτηση για τα σημεία 10, 11 και 12. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ιαπωνίας και συγκεκριμένα η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Έχουμε στην αρχή μια σύντομη παρουσίαση της αντιπροσωπείας μας που πήγε 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο. Ήταν ε, μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, ε, διερευνητική για να δούμε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ε, συμφωνία, τι γίνεται με τα θέματα της σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, πώς εφαρμόζεται και πώς κυρώνεται από την Ιαπωνία η ροή δεδομένων, διατάξεις που ισχύουν για την προστασία των καταναλωτών. Είχαμε πολύ γόνιμε συζητήσει με όλου τους ενδιαφερομένους, ενεχομένους εκεί στην Ιαπωνία, Υπουργεία. Είδαμε τον Υπουργό Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργό Εξωτερικών ε, και τον Υπουργό ε, εργασία και άλλους πολλούς ε, και τον Υφυπουργό Γεωργίας και ένα ειδικό σύμβολο του Πρωθυπουργού Άμπε. Συζητήσαμε και με ομολόγους μας βουλευτές και πάρα πολλούς ενδιαφερομένους και μεταξύ αυτών ήταν η βιομηχανία, η Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων, Κοινωνία των Πολιτών. Έχουμε μια πλήρη εικόνα της συμφωνίας αυτής. Και η κατάσταση στην Ιαπωνία ε, εν ώψη αυτής της συμφωνίας ξέρουμε πλέον ποια είναι. Εκφράσαμε και τις δικές μας επιθυμίες, την επιθυμία μας μάλλον να συνεισφέρουμε ε, στην ολοκλήρωση και υλοποίηση αυτής της συμφωνίας και τελικά νομίζω ότι ήταν χρήσιμη η επίσκεψη. Και δεν πρόκειται η κύρωση να γνωρίσει κανένα μεγάλο πρόβλημα και ούτε να έχει προβλήματα και προσκόμματα. Θα δώσω μέσα το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Πέντρο Σίλβα Περέιρα, ο οποίος ήταν και εκείνο μέλος της αντιπροσωπείας. Ρενική εισηγητής και για τις δύο συμφωνίες. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ, η αποστολή της ΣΥΝΤΑ στην Ιαπωνία ήταν επίκαιρη και πολύ επωφελής. Ε, σε τρία θέματα θα ήθελα να εστιαστώ, εν συντομία. Το πρώτο είναι ότι πέραν του ότι συναντηθήκαμε με βουλευτές, με επιχειρηματικές ενώσεις, συνδικάτα, ε, οργανισμούς καταναλωτών και ΜΚΟ, είχαμε επίσης και την ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες πολιτικές συναντήσεις ε, υψηλού επίπεδου με υπουργού, ε, το οποίο αποτελεί και πολιτικό μήνυμα της δέσμευσης της Ιαπωνίας σε αυτή την Συμφωνία εταιρική σχέση. Δεύτερον, είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε και τα δικά μα μηνύματα, κυρίω όσον αφορά τη σπουδαιότητα των δεσμεύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων, όπω αναφέρατε, των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, τη κλιματική αλλαγή, ε, τη καταπολέμηση παράνομη υλοτομία και ειδικότερα τη ανάγκη ε, κύρωση των δύο ε, από μηνασών συμβάσεων τη ILO. Στείλαμε και ένα μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι η ε, θέση σε ισχύ της συμφωνίας ε, και δεν υπήρχε καμία ένσταση. Ε, ο ειδικό σύμβουλος του Πρωθυπουργού Άμπε Δεύτερον ανακοίνωσε στην αποστολή μας ότι η Ιαπωνική κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα διυπουργικό πλαίσιο που θα ασχοληθεί με την υλοποίηση των δεσμεύσεων βιώσιμης ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης τη κύρωσης των δύο συμβάσεων του ΑΕΛΟ που απομένουν. Εμείς φυσικά ζητήσαμε συγκεκριμένα βήματα για την κύρωση και αυτό πράγματι αποτελεί ένα συγκεκριμένο βήμα προς τα εμπρός, το οποίο καλωσορίζουμε ως θετική εξέλιξη. Όσον αφορά το σχέδιο ψηφίσματος και το σχέδιο σύστασης, ε, σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα που σας έχουμε υποβάλει, ε, στο δικό μου σχέδιο ψηφίσματος και το σχέδιο σύστασής μου ε, που σας έχω παρουσιάσει για τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Όπω βλέπετε, η πρότασή μου είναι σαφή. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να δώσει την ε, κύρωσή του στην ε, συμφωνία με την Ιαπωνία. Να συμφωνήσει για την κύρωση για δύο βασικού λόγου. Πρώτον, είναι μέγιστη στρατηγική, μείζονο στρατηγική σημασία μια τέτοια συμφωνία με την Ιαπωνία. Είναι μια ισχυρή επιχειρηματική και πολιτική συμφωνία με ένα μεγάλο, ε, μια μεγάλη, πολύ σημαντική χώρα αντίκειται στην προστατευτική ατζέντα του Τραμπ, ε, υποστηρίζει το διεθνέ εμπόριο, προωθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τι ευρωπαϊκέ αξίε ε, στην περιοχή τη ε, Ασία και του Ειρηνικού. Δεύτερον, η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική οικονομικά. Παρέχει τεράστιε δυνατότητε οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη διμερή εμπορική συμφωνία που έχει κλείσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε τεράστιο στο του παγκόσμιου ΑΕΠ και του παγκόσμιου εμπορίου και αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί του εμπορίου στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Και τέλος ε, είναι μια πολύ καλά ισορροπημένη συμφωνία που υπερασπίζεται τα δικά μας συμφέροντα στην Ιαπωνική αγορά και διασφαλίζει τους ευαίσθητους τομείς μας εκ των ε, οι πιο ευαίσθητοι όπως αποδείχθηκαν στις διαπραγματευτικές ε, ε, διαδικασίες ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία, η γεωργία, όλοι αυτοί βρίσκονται μέσα στη συμφωνία. Δεύτερον, αυτή η συμφωνία ανοίξε μια νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών. Λαμβάνει υπόψη τι ανησυχίε σε θέματα βιώσιμη ανάπτυξη. Από αυτή την άποψη, σε σύγκριση με τη συμφωνία που μόλις συνάψαμε με τον Καναδά, καλό θα ήταν να πούμε ότι η παρούσα συμφωνία είναι ΣΥΤΑ Είναι μια βελτιωμένη έκδοση της ε, συμφωνίας με τον Καναδά. Αναφέρεται σαφώς και ρητά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, για πρώτη φορά περιλαμβάνει μια αναφορά στην Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, πέραν φυσικά όλων των άλλων ε, ε, πλειονομερών ομερών διεθνών συμφωνιών. Έχει μια σαφή διάταξη, ρητή διάταξη για τη βιοπικιλότητα, για την ε, ε, εταιρική ευθύνη βάσει των αρχών του ΩΣΑ. Περιλαμβάνει μια εντολή για την για το εμπόριο ε, σε επαφή και με την κοινωνία των πολιτών προωθεί τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα ε, ευρωπαϊκά, ε, ε, διεθνή πρότυπα και της Ιαπωνίας. Επίσης σημαντικό πράγμα από άψη προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον η συμφωνία αυτή υλοποιεί και τη δέσμευση προώθησης της βιώσιμης γεωργίας με μηχανισμούς συνεργασίας συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της υπαίθρου, των ανασφαλών τροφίμων για τους καταναλωτών και την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και αλίας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι 205 γεωγραφικές ενδείξεις λαμβάνουν προστασία δύναμη αυτής της συμφωνίας. Να συμφωνήσω ότι με τον Καναδά επιτύχαμε μόνο 143 ε, γεωγραφικές ενδείξεις να προστατευτούν. Οπότε δημιουργήσαμε μια κοινή συνεννόηση με την Ιαπωνία για το τι σημαίνει προστασία γεωγραφικών ενδείξεων. Όπω γνωρίζετε, η συμφωνία αυτή δεν έχει καμία αναφορά στην προστασία των επενδύσεων. Αυτή θα ακολουθήσει άλλη οδό. Δεν κάναμε αυτή τη συζήτηση, θα, το, θα την κάνουμε, δεν κάναμε καμία συζήτηση για το ISDS. Υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρηση για τι ροέ δεδομένων. Και τέλος, και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, η συμφωνία περιλαμβάνει μια ρήτρα αναθεώρησης όσον αφορά τη δυνατότητα υλοποίηση του κεφαλαίου βιώσιμη ανάπτυξη, όπω έχουμε συμπεριλάβει και στην Καναδική Συμφωνία. Αυτό όμω παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης των μηχανισμών ε, υλοποίηση ε, του κεφαλαίου βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύω θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία όσο το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, να κάνω μία αναφορά στις ε, συμβάσεις του ILO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Να πω ότι ε, υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις για την κύρωση των συμβάσεων ε, του ILO και θα πρέπει να καλωσορίσουμε το γεγονός ότι επιτέλους η Ιαπωνία προχωρά με συγκεκριμένα βήματα προς τη δημιουργία αυτού του διπουργικού πλαισίου. Αυτό είναι το σκεπτικό που στηρίζει την έγκριση αυτής της συμφωνίας. Αναμένω τα σχόλιά σα και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τους σκιώδεις ε, όσον αφορά τι τροπολογίε του, για να βελτιώσουμε την πρότασή μου. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, Πέντρο. Ευχαριστώ πολύ, Πέντρο. Θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις συζητητέ για το ΕΛΚ. Ε, ο Ντάνιελ Κασπάρη έχει το λόγο δεν είμαι ακριβώ σκιώδη εισηγητή, αλλά θα τοποθετηθώ. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε παρατηρήσει. Όπω και να έχει, νομίζω πω είναι πολύ καλό πω ε, συμφωνούμε για το ότι η συμφωνία με την ε, Ιαπωνία έχει τύχει πολύ καλή διαπραγμάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ακόμα καλύτερη από την ε, ΣΕΤΑ. Οπότε συμμερίζομαι την άποψη ότι είναι μια συμφωνία ΣΕΤΑ-ΣΥΝ, αν θέλετε. Όμως, έχω ορισμένε δυσκολίε με κάποια σημεία τα οποία ε, δείχνουν πώ ασχολούμαστε με την Ιαπωνία, πώ αντιμετωπίζουμε την Ιαπωνία. Η, η Ιαπωνία είναι μια δημοκρατία, ελεύθερη δημοκρατία για, χρόνια, για πολλά περισσότερα χρόνια από ότι ορισμένε ε, χώρε κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πω ότι με λυπεί για το, το γεγονό ότι ε, ορισμένε ε, χώρε χρησιμοποιούν την συμφωνία αυτή για να περάσουν τη δική του προσωπική ατζέντα. Να σα πω λοιπόν ότι θεωρώ αρκετά παρά τολμώ τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το, κάποια πράγματα, το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης για παράδειγμα, ε, και τον τρόπο με τον οποίο σαν να θέλουμε να διδάξουμε ε, στους Ιάπωνες. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να δείξουμε προσοχή ε, αλλά μην ξεχνάτε, η Ιαπωνία είναι μια δημοκρατία λειτουργικότατη, αντιρωσοπευτική, ε, ε, με νομοθεσία που προστατεύει τους, εργαζομένους και από την άλλη ε, βλέπω ότι αντιμετωπίζουμε την, ορισμένη μάλλον, όχι όλοι, αντιμετωπίζουν την Ιαπωνία σαν να είναι μπανανία. Είναι απίστευτο. Ζητούν αφοπλισμό, ζητούν το ένα, ζητούν το άλλο, είναι ντροπή. Ε, το πώς επιχειρηματολογούν ορισμένες ε, χώρες απέναντι στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει δικές, δική της νομοθεσία, δικές της ε, μεθόδους για να κάνει κάποια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτές τις διαφορές πρέπει να τις αναγνωρίζουμε. Επίσης τίποτα από αυτά που δεν κάνει δεν αντιβαίνει στο, διεθνέ, στο διεθνές δίκαιο. τώρα, προστασία των επενδύσεων, όπως και στην TTIP, να επαναλάβω και εδώ ότι πρόκειται για δημοκρατίες, ε, δεν χρειάζεται ε, να είμαστε υπερβολικοί. Νομίζω πως ε, στην προστασία των επενδυτών, ακριβώς όπως και στην προστασία των επενδύσεων και στον Διεθνή Οργανισμό Εργασία, Προστασία των Εργαζομένων, πρέπει να ε, αναγνωρίζουμε το γεγονό ότι η Ιαπωνία είναι δημοκρατική χώρα, επαναλαμβάνω, και δεν ε, είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακλάρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρου τη ομάδα SCR, η οποία καλωσορίζει την έκθεση αυτή και θεωρεί πω το κείμενο είναι αντιπροσωπευτικό και τονίζει τα κύρια στοιχεία τη ε, συμφωνία για τις δημόσιες προμήθειες, για τις δημόσιες υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών. Επίσης, τονίζει ότι έχει στρατηγική σημασία η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας και ε, επαναλαμβάνω, ε, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το πολυμερές ε, σύστημα δείχνει το μέλλον, δείχνει το δρόμο προς το μέλλον και θα πρωτοστατήσει στην, στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων χωρών του Ειρηνικού. Χρειάζεται όμως ε, βελτίωση, υπάρχει περιθώριο και νομίζω πως το τροπολογίες μας θα συνεισφέρουν σε αυτό. Ε, η συμφωνία θα φέρει πολλά ωφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές με την ε, κατάργηση των δασμολογικών και μη φραγμών για προϊόντα, για παράδειγμα, όπως τα φαρμακευτικά ή τα ιατροτεχνολογικά. Αυτό θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη από κεφάλαιο για να καλύψουν τις ανάγκες τους και ε, επίσης ε, θα βοηθήσει στην ανταλλαγή πληροφοριών για την πρόσβαση στην αγορά. Επίσης χαιρετίζουμε τις προτάσεις του ε, εισηγητή για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, είναι πολύ σημαντική επίσης η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μέσω συμβουλευτικών ειδικών ομάδων και ε, χρειάζεται, ορισμένα κεφάλαια χρειάζονται βελτίωση. Αυτά προς το παρόν. Αναμένουμε μια καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συνεισηγητές. Και να επαναλάβω και εγώ αυτό που είπε ο συνάδελφος Κασπάρη ότι όσοι έχουν προστατευτικές απόψεις, ας μην έχουν ψευδεστήσεις ότι οι εταίροι μας ε, είναι και αυτοί έτσι. Οι εταίροι μας αξίζουν περισσότερο σεβασμό από αυτόν που τους παρέχεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χίρς, εκ μέρου των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσο φιλελεύθερη ομάδα στηρίζουμε και εμείς την εμπορική συμφωνία με την ε, Ιαπωνία. Χαιρετίζουμε τη συμφωνία αυτή από τη μία επειδή είναι ένα ε, πολύ επίκαιρο μήνυμα για τις ε, σχέσεις μας. Είναι απόλυτα αναγκαίο λοιπόν να το στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι θέλουμε ένα ελεύθερο εμπόδιο, εμπόριο και ότι αυτό είναι δυνατό. Από την άλλη, η συμφωνία αυτή είναι στρατηγική σημασία, θα είναι ωφέλιμη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις και για την ίδια την οικονομία, ε, με ξοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ε, με την κατάργηση των ε, τελωνιακών δασμών. Επίσης, να πω πως με εξέπληξαν θετικά ε, οι εξελίξει των ε, διαπραγματεύσεων, η συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτές και η πολύ θετική στάση τη Ιαπωνία απέναντι σε όλα αυτά. Ε, φυσικά Υπήρξαν και κριτικές, οι οποίες ε, όμως ήταν θετικές και η Ιαπωνία είναι δεκτική προς αυτή την κριτική. Κάτι άλλο, ροή δεδομένων, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει πιστεύω να ενισχυθεί, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, νομίζω πως ε, εδώ θα βρούμε αποδοχή ευήκο αότα διότι πρέπει να συνεχίσουμε ε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ε, επίσης, ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ένας κανονισμός στον οποίο έχουν, έχει ασκηθεί κριτική, ιδιαίτερα μάλιστα ε, σε σχέση με την αντιμετώπιση μας με την Κίνα. Σχέση μας με την Κίνα. Νομίζω πως βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, γι' αυτό λοιπόν στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή απόλυτα 100% και σε ό,τι αφορά το ίδιο το ψήφισμα, νομίζω πω έχει πάρα πολύ καλά θετικά επιμέρου σημεία. Θα υποβάλουμε όμως ορισμένες τροπολογίες ε, για τα ε, θέματα που θέλουμε να συμπληρώσουμε. Ωστόσο, οι κυρώσει στο σημείο 11 είναι ένα σημείο με το οποίο έχουμε πρόβλημα. Νομίζουμε πω δεν είναι αυτό ο σωστό δρόμο, αλλά θα υποβάλουμε σχετικέ τροπολογίε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Κλάου Μπούχνερ, μέρο των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για, τα, για του, του. Πρέπει όμως ε, να αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν προβλήματα στη συμφωνία. Καταρχάς, ισχύει ότι η συμφωνία αυτή είναι ε, μια συμφωνία που δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στο πλαίσιο της αύξησης του προστατευτισμού που παρατηρείται. Ωστόσο, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω έχει χάσει την ευκαιρία να ξεκινήσει αλλαγές για να αλλάξει τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό στην εμπορική πολιτική ε, να παραδεχτούμε ότι το status quo δεν είναι βιώσιμο πλέον και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, συνοχή και συμφωνία με τα διάφορα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Να αναφέρω επίσης τρία βασικά θέματα. Πρώτον, το κεφάλαιο για τις υπηρεσίες. Εδώ, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα προστατεύει το δικαίωμα ε, της ε, ρύθμισης, νομοθετικής ρύθμισης. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα της ξυλίας. Πώς μπορούμε δηλαδή να επιβεβαιώσουμε ότι οι διατάξεις ε, στο ανάλογο κεφάλαιο αρκούν για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παράνομης υλοτομίας και να φροντίσουμε ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών δεν θα ε, παραβλέψει το ζήτημα αυτό. Τρίτον, μηχανισμός επιβολής ε, των, της βιώσιμης ανάπτυξης στο εμπόριο. Εδώ και πάλι υπάρχει το ίδιο θέμα με το status quo. Και η κοινωνία των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι φορεί ε, ζητούν ε, μια προσέγγιση βασισμένη σε κυρώσει. Η Ιαπωνία έχει συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο στα πλαίσια της συμφωνίας TPP. Στη συμφωνία ΣΕΤΑ βλέπουμε ότι η ρήτρα αναθεώρησης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, αυτό διότι λείπουν ορισμένα βασικά πράγματα. Γι' αυτό η Επιτροπή πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί τα κεφάλαια για την βιώσιμη ανάπτυξη του εμπορίου. Επίσης, εμείς ε, θεωρούμε πως θα μπορούσαμε να αναστείλουμε την ε, κύρωση της συμφωνίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το θέμα. Διαφορετικά το μήνυμα που θα στείλουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση και δεν επιθυμεί να αλλάξει την εμπορική της πολιτική. Και ένα σχόλιο ε, προς τον κύριο Κασπάρη και αυτά που είπε. Προσωπικά ο ίδιος ήμουν στην Ιαπωνία, εργάστηκα για ένα χρόνο και νομίζω πως ξέρω πολύ καλά πως έχει κατάσταση εκεί. Το εργατικό δίκαιο στην Ιαπωνία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα μεταβατικό στάδιο. Γίνονται αλλαγέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε και να δούμε ότι πριν από πολλά χρόνια υπήρχαν άλλες συνθήκες. Τώρα όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε, ε, να ενισχύσουμε το εμπόριο, να δούμε πώς θα ε, διαμορφωθεί το εμπόριο αυτήν την εποχή, τη σήμερα ημέρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου τη ΓΚΟ, ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζω από τα σχόλια του κυρίου Μπούχνερ προ τον κύριο Κασπάρη και θα τα πω και εγώ γερμανικά. Εμείς δεν ήμασταν τμήμα τη αντιπροσωπείας, δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε, διότι δεν μας το επέτρεψε αυτό ο συνάδελφος Δεχόντ, το σύστημα δηλαδή κατανομής των θέσεων. Εμείς όμως έχουμε επαφές και θέλουμε να είμαστε ε, υπέρ των ανταλλαγών. Έχουν έρθει και πολλές φορές οι Ιάπωνες εδώ και στο Στρασβούργο και έχουμε και επαφές ετών και με συνδικαλιστές και με βουλευτές και τα λοιπά. Και ξέρετε, έχουμε σημειώσει και εμείς ότι και στην Ιαπωνία έχουν αντιπολίτευση. Και υπάρχει δημοκρατική διαβούλευση για να καταλήξουν στη συμφωνία αυτή τη διμερή. Και αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το έχει υπόψη όταν ανταλλάσσει απόψεις ε, μεταξύ των πολιτικών ομάδων και αξιολογεί τη συμφωνία. Συνεχίζω στα αγγλικά. Για το σημείο όπου δεν έχει γίνει επαρκή διαπραγμάτευση για τη συμφωνία κατά την απόψή μας. Πρώτη, η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι πολύ ευρύ ε, το πεδίο εφαρμογής και στο παρελθόν ε, αυτά οδήγησαν σε χρηματοοικονομική κρίση και το λέω αυτό σήμερα 10 χρόνια μετά την κρίση της Lehman Brothers. Χρειάζεται και κανονιστική συνεργασία αλλά να μην είμαστε όμοιροι των ε, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ε, και στην έκθεση ε, συμπεριλαμβάνονται κάποια στοιχεία για το περιβάλλον που δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Υπάρχει συμφωνία των Παρισιών. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη γενική μας προσέγγιση στο πώς οργανώνουμε τις εμπορικές μας σχέσεις και τι σημαίνει αυτό για τη μεταφορά των αγαθών συμπεριλαμβάνεται αυτό στην τιμή παραγωγής, ε, στη διαμόρφωση της τιμής ε, των προϊόντων που κυκλοφορούν με βάση τη μερή συμφωνία ανά την υφήλιο. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία για το περιβάλλον που δεν υπάρχουν στο κεφάλαιο του ε, περιβάλλοντος. Έχουμε επαφές λοιπόν με οι Ιάπωνες οι οποίοι τι μας λέγουν. Ότι η συμφωνία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά Ε, την ε, ξυλία και την υλοτομία γιατί θα προωθηθεί η ε, λαθρέα υλοτόμηση καθώς καταργούνται όλοι οι δασμοί στα προϊόντα ξυλίας. Σε ό,τι αφορά την αλία θα πρέπει να σταματήσει αμέσως η εμπορική φαλενοθυρία. Επίσης, ένα είδος τόνου κινδυνεύει με εξαφάνιση από την υπεραλίευση. Ε, θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να τα σκεφτεί όλα αυτά και να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Και στη συνέχεια η Ιαπωνία ακόμα δεν έχει κυρώσει ε, την ε, συμφωνία ILO που ανέφερε ο κύριος Μπούχνερ του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και θα πρέπει να βάλουμε στην έκθεση και το προτείνουμε και προς τον εισηγητή αυτό ορισμένα θέματα που θέλουμε να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ε, Συμβούλιο για τη ροή δεδομένων, τους του κανονισμούς κτλ. Η κυρία Μπεγκίν από την FTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Δεν θα έλεγα ότι συμφωνώ 100% με το κείμενο τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Δεν μπορώ να δεχθώ εύκολα κάποια σημεία. Αλλά αφού έγινε έκκληση να το δεχτούμε ή να την απορρίψουμε, στο σύνολο πρέπει να πω ότι συμφωνούμε με την ε, συμφωνία αυτή. Η Ιταλία έχει τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα με την Ιαπωνία. Εξάγουμε πολλά περισσότερα από ό,τι εισάγουμε κάθε χρόνο και το ίδιο ισχύει για πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Είμαι βέβαιη λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή θα είναι επωφελή ε, και για τι Ιταλικέ και για τι ε, επιχειρήσει των υπόλοιπων χωρών και για του πολίτε μα. Συμφωνούμε με τα όσα έγιναν για τι δημοσιογορέ. Ζητήσαμε απόσυρση κάθε δασμού για τα γεωργικά προϊόντα από την Ευρώπη, τα οποία εξαγαγούμε τώρα στη χώρα των ατέλων του Σιλίου χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, αξιολογώντας συνολικά, δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποιε συγκεκριμένε πτυχέ που δεν μα έχουν πείσει. Αντιτίθεμε σαφώ ε, στην ε, αρνητική λίστα όσον αφορά το κεφάλαιο για τις υπηρεσίες σε ορισμένα άρθρα του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και διαμαρτύρομαι διότι η Ιαπωνία δεν έχει κυρώσει όλες τις ε, συμβάσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Χαίρομαι ωστόσο που δεν έχει ληφθεί υπόψη η ρήτρα STS ή SDS στο συμφωνία αυτή. Θα ήθελα να αποτρέψω την Κομισιόν από την ιδέα το να συμπεριλάβει τέτοιου μηχανισμού και στο μέλλον. Ουδέποτε θα συμφωνήσουμε εμεί σε ε, συμφωνίε τέτοιε με ανεπτυγμένε χώρε. Η Ιαπωνία είναι μια από τι πλουσιότερε χώρε του κόσμου. Έχει τεράστιε δυνατότητε ε, ε, οικονομικές και επιθυμία αγοράς προϊόντων ποιότητας Ιταλικών και Ευρωπαϊκών. Με αυτή τη συμφωνία θα βοηθήσουμε λοιπόν και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Τιτσιάνα και για το ΙΕΝΕΦ, e η κυρία Ζαμέ. Ε, ευχαριστώ. Εγώ δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας, λέει η κυρία Ζαμέ. Ε, ε είναι σαν μια συμφωνία ΣΕΤΑ ε, ΣΥΝ. Ναι, αλλά ποιο θα διαπραγματεύτηκε αυτά, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο κύριο Γιούγκερ Αφορά το 1 τρίτο του παγκοσμίου ΑΕΠ, 40% ε, των συναλλαγών των παγκοσμίων και 600 εκατομμύρια καταναλωτέ. Και εμεί είμαστε η τρίτη εμπορική εταίρη τη Ιαπωνία. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε εμεί ότι θα πρέπει κάθε εθνικό κοινοβούλιο να κυρώσει τη συμφωνία, πράγμα που δεν γίνεται. Επίση, ε, δεν έχουν οριστεί ε, τα, των διακανονισμών και τη διαιτησία είναι επικίνδυνο αυτό. Επίσης ε, μιλάτε για την προστασία 205 ονομασίες προέλευσης από τα 1534 προϊόντα σταγόνα στον ωκεανό. Εντάξει, υπάρχει η φαλαινοθυρία Υπάρχει το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που ε, προχωράει πάρα πολύ σε εμά και οι Ιάπωνες θα έρθουν να μας κατακλείσουν με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και έχουμε και άλλα θέματα, ε, ε, ζωικά προϊόντα, βόλιο, κρέας, χείριο κρέας, χοιρινό. Τρώνε τέτοια πράγματα οι Ιαπωνέζοι κάθε μέρα. Ε, δεν είναι φαλαινοθυρία. Υπάρχει ο κόκκινο τόνο, ε, βιομηχανική αλεία, η Ιαπωνέζικη, η οποία ε, στη Μεσόγειο έχει ρημάξει τα πάντα. Δεν ενδιαφέρονται για τη διαφύλαξη των ειδών, αλωνίζουν. Φέρνουν εργοστάσια στη Γαλλία που ρηπαίνουν αυτή η συμφωνία που είναι πραγματικά τεράστια και έχει τρομακτικές συνέπειες ε, ε, και απειλεί επικίνδυνα την απασχόληση της βιομηχανίας μας και τα λοιπά και για να μην μιλήσω και για την ε, υγεία του καταναλωτή και σε σχέση με τη ΣΕΤΑ. Μιλάμε για προστασία. Ε, εγώ θέλω μια ασπίδα που να προστατεύει. Μόλις ακουστεί η λέξη εδώ προστατευτισμός, εξαγριώνεστε. Δεν είναι καλό πράγμα οι ελεύθερε συναλλαγέ. Καλά θα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα να προστατεύει τα ευρωπαϊκά έθνη και μετά να ανησυχεί για τι ε, πολιεθνικέ και τι παγκόσμιες business. Θέλω να επανέλθω σε Κάτι που μάθαμε μέσα στη νύχτα. Ο κύριος Τραμπ ε, που καφιέστε ότι έχετε καταλάβει την ε, προστατευτική του ατζέντα, ε, θα συμφωνήσει με τους Ιάπωνες. Και σε ποιο θα στραφεί η Ιαπωνία τώρα, προς τις Ηνωμένε Πολιτείες, αφού καταλήξει η συμφωνία μαζί μας. Λοιπόν, Υπάρχει ο τύπος και η ουσία. Κάποια στιγμή, λυπάμαι πάρα πολύ, θα πρέπει να ε, μιλήσουμε και για ε, ακύρωση αυτών των συμφωνιών. Και κύριε Κασπάρη, δεν θα πρέπει να διδάξουμε στην Ιαπωνία Δημοκρατία, αλλά στην Κομισιόν και στον κύριο Γιούνκερ τους κανόνες της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκαν εδώ οι σκιώδεις εισηγητές. Και τώρα, λυπάμαι μέλη της Επιτροπής, έχω πολλούς που ζητούν το λόγο. Θα σας περιορίσω το χρόνο γόρευσης. 1,5 λεπτό έκαστος. Hansen. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ εκπροσωπώ τη σχεδή ηγετρία σήμερα του ΕΛΚ που ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ε, τον εισηγητή του ΕΛΚ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεση και για τη σύσταση. Δεν έχω σχόλια. Κάνετε πολύ καλή δουλειά, κύριε Σίγητα. Υποστηρίζω τη βάση της έκθεσης, αλλά θέλω να σχολιάσω δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, υπογραμμίζουμε ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, το ΑΕΠ, οι θέσει εργασία και ανάπτυξη χάρη σε αυτή τη συμφωνία. Επίση, να τονίσουμε ότι είναι σημαντική εξαγωγική αγορά για του Ευρωπαίου γεωργού, η Ιαπωνία και για του παραγωγού τροφίμων. Καλωσορίζουμε λοιπόν τι αυξημένε εξαγωγικέ δυνατότητε που παρέχει η συμφωνία για τα αγροδιατροφικά προϊόντα μα. Επίσης, η συμφωνία θα διευκολύνει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες ε, στην πολύ ευρεία η Ιαπωνική αγορά. Θα βοηθήσει αυτό το εμπόριο υπηρεσιών μα. Εμεί θα υποβάλουμε σχετικέ τροπολογίε. Ανέκαθεν μιλούσα υπέρ μια εταιρική σχέση μεταξύ, μεταξύ Ιαπωνία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενισχύσει το εμπόριο σε προϊόντα και υπηρεσίε και θα αυξήσει τι ευκαιρίε ε, επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία. Πιστεύω τώρα ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει το ταχύτερο δυνατόν την έγκρισή του σε αυτή τη συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε να εστιαστούμε στην υλοποίηση τη εμπορική αυτή συμφωνία ούτως ώστε όλοι να επωφεληθούν από αυτήν. Ευχαριστώ. Και τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις από εξ μου, γιατί και εγώ συμμετείχα στην αποστολή στην Ιαπωνία, η οποία είχε θετική έκβαση. Μας δεχθήκαν οι ομολόγοι μας με μεγάλο ενθουσιασμό εκεί, όχι μόνο εξωματούχοι, αλλά από υπουργεία, αλλά και τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Συναντηθήκαμε με την Ένωση Καταναλωτών, τη Συνεταιριστική Ένωση των Καταναλωτών, ακόμη και η κοινωνία των πολιτών δηλαδή στην Ιαπωνία γνωρίζει πολύ καλά τι ε, αποτελέσματα και ωφέλη θα έχει αυτή η συμφωνία για ολόκληρη τη χώρα και για την κοινωνία των πολιτών. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε κάποια πολύ αυτά παραδείγματα μάλιστα, ότι η Ιαπωνία καταβάλει προσπάθειες κύρωσης ε, των δύο συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας που απομένουν. Φέτος είχαμε την πρώτη αναθεώρηση τη εργασιακή νομοθεσία στην Ιαπωνία μετά από 70 χρόνια. Αυτό αποτελεί ένα καθαρό μήνυμα ότι η Ιαπωνία προχωρά. Σω να μην πηγαίνουν όλα τέλεια. Ε, ε ίσως και εμεί να μην προχωράμε τόσο γρήγορα. Πρέπει όμω να παραδεχτούμε ότι κάνουν βήματα προ τα εμπρό. Έχουμε κάνει και άλλε συμφωνίε με λιγότερο προοδευτικού εταίρου. Οπότε πραγματικά πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αυτή την ειλικρίνεια από πλευρά τη Ιαπωνία. Είναι καλό σήμα για να προχωρήσουμε μπροστά και θα πρέπει να αποφύγουμε να αναφέρουμε κυρώσει και τέτοια πράγματα στο ψήφισμά μα. Όταν αναφέρουμε κυρώσει, δεν μπορούν να μα πάρουν τόσο σοβαρά τέτοια εταίροι. Πρέπει να το αποφύγουμε. Στην Ιαπωνία επικυρώσαμε το, την πρόθεσή μας να έχουμε την ψηφοφορία στην Ίντα το Νοέμβριο και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό, πιστεύω, και από πλευρά μου δεν έχω παρα... ελάχιστε παρατηρήσει όσον αφορά την έκθεση του εισηγητή, που είναι εξαιρετική. Απλά για τα σημεία 10 και 11 θα, κάνω, θα υποβάλω κάποιε τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκράφαλτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία μπορεί να δώσει κίνηση στην ανάπτυξη και να σας θυμίσω ότι είχαμε παρόμοια άποψη για διάφορα άλλα θέματα για μηχανισμό επιβολή κυρώσεων, για παράδειγμα, τους οποίου έχουμε υπερψηφίσει. Βέβαια, τώρα εν ώψη προεκλογικού αγώνα υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, έχουν αλλάξει οι γνώμες, όμως ε, νομίζω πως αν πρέπει να συζητηθεί ε, κάτι, καλύτερα να γίνει ουσιαστική συζήτηση, όχι απλά να ε, είμαστε τόσο απόλυτοι. Η Ιαπωνία είναι μια αναπτυγμένη χώρα η οποία δεν έχει κερδίσει τέτοια ε, αντιμετώπιση. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω πως ε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όταν συζητάμε έτσι. Νομίζω πως η πρόταση δεν είναι τόσο φιλόδοξη όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Επίσης οι μηχανισμοί επιβολής δεν προβλέπονται στο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα και για το εμπόριο. Επίση, σε ρήτρα αναθεώρηση, ε, η, Ιαπωνία δεν έχει δείξει τέτοια φιλοδοξία. Αυτό το έχουν δείξει οι συνομιλίες που είχαν οι συνάδελφοί μα με την Ιαπωνική πλευρά και νομίζω πω είναι ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, διότι χρειάζεται ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων ε, και να έχουμε δυνατότητα αντίδραση σε περίπτωση παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών. Μετά ε, πρέπει να επενέσουμε ορισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει από την Ιαπωνική πλευρά, όμως να ξέρετε πως ε, οι πολίτε, η κοινωνία των πολιτών της Ιαπωνίας δεν είναι τόσο κινητοποιημένη όσο εμείς, γι' αυτό χρειάζονται ακόμα προσπάθειες. Η, η Ιαπωνία χρησιμοποιεί μία επιστημονική ε, προσέγγιση και αυτό διαφέρει από την, ε, τις δικές μας ε, μεθόδους. Δεν έχουμε πρόβλημα με το εμπόριο, έχουμε πρόβλημα με το μη ρυθμισμένο εμπόριο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρασφαντερή. Ο κύριος Σάινφελτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να στηρίξω και εγώ την άποψη του κύριου Κασπάρη. Συμμερίζομαι τις απόψεις του και πραγματικά νομίζω πως είναι αποθητικό να ακούς ε, απόψεις που δεν ασκούν κριτική στην ε, η Ιαπωνία, πως ασκούν κριτική σε έγγραφα τα οποία δεν έχουμε στην ολότητά τους. Ε, με αποθούν αυτά τα σχόλια του να μην ε, κυρώσουμε τη συμφωνία, του να αναστείλουμε τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι υποδειγματική θα έλεγα. Ίσως η καλύτερη που είχαμε μέχρι τώρα ανάμεσα σε όλες αυτές τις συμφωνίες που έχει κυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα. Η Ιαπωνία ως εταίρος μας κατά την άποψή μου είναι ένας σημαντικότατος εταίρος ο οποίος έχει υπόβαθρο, πολιτισμικό, εμπορικό. Έχει μεγάλη ιστορία. Βέβαια, όλα αυτά ε, δεν έχουν τόσο σημασία. Να πω κλείνοντας ότι σε ό,τι αφορά τον ε, τα εργασιακά δικαιώματα, ε, να σας ε, ενημερώσω ότι οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν πολύ θετική άποψη για τα όσα συμβαίνουν στην Ιαπωνία για την νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι λοιπόν πρέπει να ψάχνουμε προβλήματα στις Βρυξέλλες όταν δεν τα έχουν εντοπίσει οι ειδικοί. Ευχαριστώ, Εμμανουέλ Μογέλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν ακούω τα επιχειρήματα κάποιων συναδέλφων, ενοχλούμε λίγο. Όταν ε, ε, επικρίνουμε την ε, άκρατη τη συναλλαγή, μας προσάπτουν ότι είμαστε τραμπικοί, είμαστε του προστατευτισμού. Ε, γιατί τέτοια χαλήνωτη χαρά και ενθουσιασμός. Εκφράζουμε επικρίσεις για κάποια πράγματα. Α, λέτε, θα μας, ε, μας λένε, θα δείτε, το Τζέφτα με την Ιαπωνία είναι ένα σέτα συν. Εγώ ανησυχώ, γιατί ε, το Ίδρυμα του Λό και άλλε περιβαλλοντικές οργανώσεις μας λένε τι έχει γίνει με τη ΣΕΤΑ και δεν είναι ενθαρρυντικά. Για τη συμφωνία αυτή υπάρχουν πολλά επιχειρήματα γεωπολιτικής φύσης. Μας λένε ότι η Ιαπωνία, εταίρος μας, δημοκρατική χώρα. Ωραία, τα ξέρουμε όλα αυτά. Τα οικονομικά επιχειρήματα όμως είναι πολύ λίγα. Και η μελέτη αντικτύπου που έκανε τον Ιούνιο το 2008 η ε, Κομισιόν έχει ενδιαφέρον γιατί λέει ότι το 2035 θα κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 0,14% του ΕΕΠ. Σιγά την επανάσταση. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ανισορροπία οποία ε, ε, ε, θα είναι ο, ο μέγας νικητής η αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας κυρίως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αναφυσβήτητο και πολύ ανησυχητικό για την ομάδα μας που θέλουμε να υπάρχει έλεγχο των τραπεζών. Ε, Παγκόσμιο Οργανισμό εργασία. Ε, υποτίθεται ότι κάναμε μια συμφωνία, αλλά είναι οφθαλμαπάτη για τα δημόσια έργα και τι δημόσιε προμήθειε, Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε επικριτικοί. Ευχαριστώ κυρία Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σα κάνει έκπληξη αυτό που θα πω, αλλά εγώ θεωρώ ότι η άπονε είναι πραγματικά κάτι το εξαιρετικό. Είναι δυνατότεροι από εμά. Όταν διαβάζει κανεί τη Συμφωνία Τζέφτα και ειδικότερα όσον αφορά τι υπηρεσίε, στον αρνητικό κατάλογο της απελευθέρωσης των υπηρεσιών, όπως τον ονομάζουμε, ήταν πιο προληπτικοί οι Ιάπωνες. Προστάτευσαν κάποια θέματα, κάποιες υπηρεσίες ε, από την απελευθέρωση που εμείς ήμασταν έτοιμοι να απελευθερώσουμε. Η Ιαπωνία είναι μια δημοκρατία ίσως και πιο προχωρημένη από την Ευρωπαϊκή από τις ευρωπαϊκές, διότι όταν λαμβάνει μια θέση το, η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, ο κόσμος τη σέβεται. Αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε υιοθετήσει διάφορες διατάξεις όσον αφορά, στο εδώ στο Κοινοβούλιο όσον αφορά μία υποχρεωτική λογική επιμέλεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδέποτε ε, εμφανίζεται, εμφανίζεται τέτοια πρόταση όταν διαπραγματεύεται διμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες. Συστηματικά τα κάνει όλα εθελοντικά. Το Κοινοβούλιο ωστόσο έχει πει Θυμάστε όταν συζητήσαμε για τα ε, ορυκτά από περιοχές σειράξεων είχε πει η Κομισιόν εθελοντικά και εμεί εδώ με μεγάλη πλειοψηφία είχαμε ζητήσει υποχρεωτική διαδικασία την οποία δεν υπερασπίζεται η Κομισιόν. Ωστόσο η Ιαπωνία στην ε, Συμφωνία του Ειρηνικού έχει συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη με κυρώσει. Και αυτό που με λυπεί εμένα εδώ δεν είναι η θέση τη Ιαπωνία αλλά η αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαπραγματευτικά και η έλλειψη σεβασμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι Δημοκρατικέ Αρχέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά και την πρόοδο που έχει επιτύχει. Γενικά πιστεύω ότι είναι καλή η συμφωνία όσο και απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεωπολιτική λόγη είναι πολύ σημαντική. Επίσης θα πρέπει να κάνουν περισσότερα βήματα η Ιαπωνία ε, στη δέσμευση που έχει αναλάβει να κυρώσει τις δύο συμβάσεις στο ΕΛΟ που εκκρεμούν. Η Διευπουργική ε, Επιτροπή έχει συσταθεί για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά χρειάζεται πραγματικά ε, κάποια συγκεκριμένη δράση. Θέλω να πω δύο πράγματα στον εισηγητή. Θα μπορούσαμε να εντάξουμε στο ψήφισμα στην έκθεσή του τον κοινό ρόλο που διαδραματίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία ε, ήδη στους διεθνείς οργανισμούς για να ε, υπερασπίζονται το εμπόριο που να βασίζεται σε κανόνες, το αντίθετο δηλαδή του Τόναλτ Τραμπ, και σε ό,τι αφορά επίσης τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ε, προασπίζεται Ε, την πολυμερή ε, συνεργασία. Κρίμα που δεν έχουμε τίποτα για τη διάσταση του φύλου. Θυμίζω ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε ε, με μεγάλη πλειοψηφία τη σχετική έκθεση για το διάσταση του φύλου στο εμπόριο. Ξέρω ότι έχει δυσκολίες η ιαπωνική κοινωνία, αλλά η αναθεώρηση του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη χρειάζεται να κάνουμε μια προσπάθεια για να προχωρήσουμε και προς την κατεύθυνση αυτή. ευχαριστώ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Λουίς Πορτέρο. Ε, thank you, Chairman. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι έλαβαν το λόγο για τη στήριξη που έδειξαν για την κύρωση της ε, συμφωνίας με την Ιαπωνία. Πολλά ήδη έχουν ακουστεί, έχουν υποθεί για τα οικονομικά ωφέλη της συμφωνίας, για την παγκόσμια σημασία αυτή και για τι συγκεκριμένε επιμέρους πτυχέ τη. οπότε δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά. Αλλά θα ήθελα να πω ε, κάτι για τη διαδικασία κύρωση τη συμφωνία. Ε, όπως γνωρίζετε ως μέλη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, η Βουλή της Ιαπωνίας επιθυμεί να κυρώσει τη συμφωνία κατά πάσα πιθανότητα τον Νοέμβριο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει και εκείνο σύντομα μετά το Νοέμβριο έτσι ώστε να ε, τεθεί σε ισχύ νωρί η συμφωνία. Αυτή η θέση σε ισχύ είναι πολύ σημαντική για διάφορους λόγους. Ένας από αυτού ίσως ο πιο σημαντικός και πιο προφανής, είναι ότι θα εξαφανιστούν πολλοί εισαγωγικοί δασμοί με την ε, θέση ισχύ της συμφωνίας. Για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά κρασιά αυτή τη στιγμή έχουν 15% δασμού ε, εισαγωγή στην Ιαπωνία. Αυτοί θα εκλείψουν, θα καταργηθούν με τη θέση ισχύ τη συμφωνίας. Είναι δηλαδή πολύ συγκεκριμένες δαπάνε τι οποίες έχουν να καταβάλουν οι επιχειρήσει και ε, μόνο να υποφεληθούν έχουν με τη θέση σε ισχύ τη ε, συμφωνίας στην Ιαπωνία. Επίσης, να σχολιάσω την δημιουργία διπουργικής ομάδας στην Ιαπωνία η οποία θα ε, μελετήσει τα κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης και εμπορίου της συμφωνίας. Ε, αυτή η ομάδα έχει συσταθεί, είναι πραγματικότητα από ό,τι ε, μου είπαν οι ιαπωνικέ αρχές έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί μας και σκοπεύουν να ξεκινήσουν έναν τεχνικό διάλογο ήδη το μήνα που μας έρχεται έτσι ώστε να δρομολογείται η συμφωνία. Αυτό δείχνει τη δέσμευση από τη δική τους πλευρά για τα κεφάλαια αυτά και για την ε, υλοποίησή τους προτού ακόμα γίνει οποιοδήποτε βήμα προς ακύρωση της συμφωνίας. Παίρνει λοιπόν η Ιαπωνία τα πράγματα πολύ στα σοβαρά, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στην αντιμετώπιση πολλών ε, ζητημάτων. Πέρυσι ε, ψήφισε νομοθεσία για την παράνομη υλοτομία, την αντιμετώπιση της, ε, προσπαθεί να χτίσει πάνω σε αυτά που ήδη έχει ξεκινήσει να φτιάχνει έτσι ώστε να αποκομίσουμε όλοι περισσότερα ωφέλη. Τέλος, κάποια σχόλια από της ουσίας και προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Να πω ότι καταρχάς παράνομη υλοτομία Ακούστηκε ότι η συμφωνία θα παροτρύνει την ε, παράνομη υλοτομία και τον πόριό τη λόγω τη απελευθέρωση των δασμών κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει νομοθεσία που έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο, η οποία απαγορεύει ε, την ε, είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά ε, προϊόντων παράνομης υλοτομίας. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως αρνητικός αντίκτυπος, καμία απολύτως ανησυχία για κάτι τέτοιο. Η συνεργασία μας με την Ιαπωνία είναι άριστη στον τομέα αυτό. Έπειτα, φαλαινοθυρία είναι προφανώς και ένα λεπτό θέμα για την Ιαπωνία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ε, τα γεγονότα τι μας λένε. Η εμπορική φαλαινοθυρία έχει ανασταλεί από το 1986 ε, βάσει της συμφωνίας της ε, Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθυρίας. Αυτό φυσικά είναι λεπτό θέμα. Ελπίζουμε να εμβαθύνουμε τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις μας με την Ιαπωνική πλευρά και να ακουστούν οι περιβαλλοντικές μας ανησυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όλους σας για τα καλά σας λόγια και για τη στήριξη που δείξατε. Επιτρέψτε μου κάποια τελικά σχόλια. Φυσικά και σεβόμαστε το κυριαρχικό δικαίωμα της ε, Ιαπωνίας ε, στην ε, νομοθεσία, αλλά θέλουμε και να ενισχυθεί η συνεργασία μας στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι σημαντικό για πολλά θέματα, για πολλούς τομείς ε, και για τη σύμβαση της ε, διεθνή οργάνωση εργασία και να σα υπενθυμίσω ότι έχουν συμπεριληφθεί παρόμοιες πολιτικές δεσμεύσει στη συμφωνία με τον Καναδά και αυτές έκαναν τη διαφορά διότι ο Καναδάς ακύρωσε τις έκρεμούσες ε, συμφωνίες της Παγκόσμια Οργάνωσης εργασία. και αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση της Ιαπωνίας χωρίς να το οποιοδήποτε κυριαρχικό τη δικαίωμα. Έπειτα, κυρώσει, Η προσέγγιση βασισμένη στις κυρώσει μάλλον. Σε ό,τι αφορά αυτές, ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με τη μελλοντική χρήση της ρήτρα αναθεώρησης. Άρα δεν συμπεριλαμβάνεται στην ε, παρούσα συμφωνία, Όμω, ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κρατήσει την ίδια θέση για την προσέγγιση βασμένη σε κυρώσει και να σα υπενθυμίσω ότι στην περίπτωση αυτή οι κυρώσει αυτέ θα εφαρμόζονται και στα δύο μέρη. Δεν είναι λοιπόν μόνο η, η που τιμωρείται, που απειλείται, οι μηχανισμοί κυρώσεων θα εφαρμόζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. διότι πρέπει να επιβληθούν και να εφαρμοστούν οι διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτοί βέβαια οι μηχανισμοί θα είναι ε, η τελευταία λύση. Τώρα, όπως ήδη ακούσαμε, η εισαγωγή παράνομης υλοτομίας ε, θα συνεχίσει να μην επιτρέπεται, θα συνεχίσει να είναι παράνομη και έχει συσταθεί μια πλατφόρμα διαλόγου που θα ενισχύσει τη συνεργασία μας ε, στον τομέα αυτό και με την Απονία και με διεθνείς οργανισμούς. Έπειτα να σας πω πως αυτή τη συμφωνία δεν κάνουμε μόνοι μας, με τον εαυτό μας. Υπάρχει πολύ θετικός κατάλογος υπηρεσιών και οφείλω να παραδεχτώ ότι το δικαίωμα νομοθε... Σίας προβλέπεται και στον τομέα των υπηρεσιών. Οι δημόσιες υπηρεσίες προστατεύονται. Δεν βλέπω να υπονομεύονται τα δικαιώματα αυτά από τη συμφωνία. Αυτά θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε, να συμπεριλάβω τις τροπολογίες σας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 2 Οκτωβρίου, 6 ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο 13 να σας ε, θυμίσω ότι απομένουν τρία σημεία στην ημερήσια διάταξη και ότι πρέπει να τελειώσουμε ακριβώς στις 12.30. Σας εκλυπαρώ λοιπόν, μην μιλάτε πολύ, να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι. Πάμε στο σημείο 13. ΠΟΕ μελλοντική πορεία. Νομίζω ότι πλέον είναι σαφές εδώ ως πρόεδρος ε, στρέφομαι προς τον εισηγητή. Αποκτώ το ρόλο εισηγητή πλέον. Για πολύ καιρό ο ΠΟΕ θεωρήθηκε ο δεδομένο ως ε, διεθνής οργανισμός. Ε, θεωρήθηκε ότι δεν ήταν πολύ δυναμικός, πολύ γρήγορος, αλλά ότι λειτουργούσε δεδομένων των αλλαγών παγκοσμίων και της στάσης των ΗΠΑ και κάποιων άλλων, θεωρώ ότι αιτιολογείται απόλυτα ή μάλιστα είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Όλοι πιστεύω κατανοούν απόλυτα ότι αυτός ο οργανισμός είναι απολύτως αναγκαίος για να έχουμε ένα παγκόσμιο εμπορικό σύστημα βάσει κανόνων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για το εμπόριο, αλλά και για άλλα θέματα. Μετά από την τελευταία ανταλλαγή απόψεών μας ε, τέλη Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δική της πρόταση για κάποιες μεταρρυθμίσεις στον ΠΟΕ. Οι προτάσεις της Κομισιόν συζητήθηκαν ε, πριν από λίγες ημέρες ε, στη Γενέβη. Συζητηθήκαν επίση και σε μια συνάντηση στην Οτάβα τέλη Οκτωβρίου. Θα συζητηθούν, συγγνώμη. Αυτή η συνάντηση έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι από τη μία πλευρά ο Καναδάς θέλει να μεταρρυθμίσουμε τον ΠΟΕ, αλλά στη συνάντηση αυτή επίσης θα υπάρχει και συμμετοχή της Βραζιλίας και της Κένιας. Όχι μόνο δηλαδή η συνήθιση ύποπτη γύρω από το τραπέζι, αλλά και κάποιες άλλες δυνάμεις. Αυτό ίσως να δώσει και μια μεγαλύτερη όθηση στη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Στη δική μας ε, έκθεση του κυρίου Ρούμπιχ και τη δική μου, κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν της Κομισιόν, προτείνοντας συγκεκριμένε προτάσει ε, μεταρρύθμιση. Μετά από την ίδρυση του ΠΟΕ, το 1959 υπήρξαν κάποια νέα στοιχεία εμπορικής πολιτικής όπως είναι σαφές. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε τώρα τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού. Γίνεται συζήτηση για ε, τη σχέση του εμπορίου με τα περιβάλλον και με τα εργασιακά δικαιώματα και τα σχετικά θεματολόγια. Αυτά πρέπει να αναγνωριστούν στον ΠΟΕ. Και στους τρεις πυλώνες λοιπόν του ΠΟΕ πιστεύω χρειαζόμαστε κάποια μεταρρύθμιση. Ε, για το βιβλίο κανόνων φυσικά, το ζήτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου, επίσης είναι ένα γνωστό ζήτημα. Υπάρχει το ζήτημα του ψηφιακού εμπορίου της ε, χειραφέτησης των γυναικών και ε, χρειάζονται κάποιοι επιπλέον κανόνες για όλα αυτά τα θέματα. Επίσης θα πρέπει ο ΠΟΕ να λειτουργεί πιο διαφανώς στο ανώτερο σώμα του, να ε, υπάρχει ένα πιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και ενδεχομένως και κάποιοι σαφέστεροι κανόνες ώστε να ληφθούν υπόψη κάποιες επικρίσεις που γίνονται και να μεταρρυθμιστεί σχετικά το ανώτερο του σώμα. Όσον αφορά την εσωτερική του οργάνωση, θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες περισσότερες ε, ε, δυνατότητες στη γραμματεία του ΠΟΕ ώστε να προωθεί ε, εργασίες του ΠΟΕ να γίνονται κάποιες προτάσεις ε, από τον ίδιο τον ΠΟΕ και όχι να περιμένουμε ε, τις προτάσεις των κρατών μελών. Στην έκθεση επίσης ε, γίνονται και κάποιες προτάσεις μεταρρύθμισης των μεθόδων εργασίας. Οπότε τίθε το ζήτημα της σταδιακής εισαγωγή μια διαφορετική προσέγγιση από την προσέγγιση της, του ενιαίου εγχειρήματο Αυτό ξεκίνησε κάπου στον Buenos Aires, ε, αν δεν κάνω λάθος. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια ευκαιρία να υπάρχει μια σαφής ρήτρα MFN ώστε να υπάρξει σαφής εταιρική σχέση. Θέλουμε επίσης και μεγαλύτερη υποστήριξη της ε, ανάπτυξης ικανοτήτων ε, με τους εμπορικούς εταίρους ώστε να μπορούν να ε, ικανοποιούν τις απαιτήσει των νέων κανόνων και να έχουν οι νεαιτέροι μεγαλύτερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στη κοινά εγχειρήματα. Αυτά είναι κάποιες σκέψεις για τον ΠΟΕ και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις μεταρρυθμιστικές. Αυτά θα βρείτε στην έκθεσή μας. Την έκθεση δική μου και του κυρίου Ρούμπιχ, ο οποίος δυστυχώς δεν ε, μπόρεσε να βρίσκεται εδώ, αλλά τον αντικαθιστώ ο κύριος Χάντσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τώρα ε, είμαι σκιώδης ε, εισηγητής, εκπροσωπώ τους σκιώδης εισηγητές του ΕΛΚ και τον κύριο Ρούμπικ. Όλο και περισσότερο ε, ζούμε σε καιρού ε, προστατευτισμού, γι' αυτό χρειάζονται σαφείς κανόνες στο εμπόριο. Η μεταξέλιξη του ΠΟΕ είναι πάρα πολύ σημαντική από πλευράς αναπτυσσομένων χωρών Τίτε πάντα η εφαρμογή των κανόνων της Συμφωνίας της Δόχα. Εμείς έχουμε ε, νέα θέματα, διαφάνεια στις ε, επενδύσεις, χρηματοπιστωτικά υπηρεσίες και άλλα. Υπάρχουν και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ε, του ΟΗΕ και οι νέες δυνατότητες της ραγδαίας ανάπτυξης της ψηφιακής αλλαγής. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να προτιμάσουμε ε, τα αναπτυσσόμενα κράτη. Aid for trade είναι το σύνθημα, δηλαδή βοήθεια με σκοπό το εμπόριο. Και στην ψηφιακή εποχή αξίζει να υποστηριχθεί. Σε ό,τι αφορά τη θεσμική μετεξέλιξη, Υπάρχει μια εμπλοκή ε, στον ΠΟΕ γιατί το σύστημα που ισχύει είναι η συνένεση. Ε, ε, υπάρχουν όμως χώρες που θέλουν να προχωρήσουν, δεν μπορεί να εμποδίζονται αυτές και οι χώρες που δεν θέλουν να συμμετέχουν από την αρχή θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε κάποια απότερη χρονική στιγμή να ενταχθούν στη συνεργασία. Για να είναι αποτελεσματικός και ισχυρός αυτός ο οργανισμός χρειάζεται πόρους και οικονομικούς και κυρίως ανθρώπινους. Γι' αυτό ε, ε, το σκοπό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και ιδιαίτερα να ενισχύσει έτσι περαιτέρω την κοινοβουλευτική διάσταση. Και τελευταίο, χωρίς να είναι το λιγότερο σημαντικό, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που ήταν και εκείνο στην πρωτοβουλία του να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ. Και το πάνελ χρειάζεται ενίσχυση για την επίλυση των διαφορών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν βάλει βέτο και δεν διορίζουν εκεί τα μέλη όμω του διαιτητικού αυτού οργάνου, ε, του δικαστέ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό οι διάφοροι σκιώδει ηγητέ, η κυρία Έμα Μακλάρκιν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, δύο συνεισηγητέ για την ε, πολύ καλή εικόνα που μας έδωσαν για το όραμά του για τον ΠΟΕ. Ε, ταυτόχρονα ως ε, μέλη του ΠΟΕ συζητούμε εδώ το ε, έγγραφο θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εξυγχρονισμό του ΠΟΕ. Το έγγραφο αυτό παρέχει λογικές λύσεις για διάφορα θέματα, για απελευθέρωση του αμπεωρίου, τονίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν ιδιαίτερα στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών και τις τα προβλήματα της μη τη μη αποτελεσματική τήρηση των ε, κανόνων του ΠΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Η... Στηρίζει την κοινή δήλωση, την τριμερή Ηνωμένων Πολιτειών ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία, αλλά θεωρώ πω θα πρέπει να γίνουν ορισμένε προσθήκε. Καταρχά, να καταστεί σαφέ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε μόνο μερό επέβαλαν ε, δασμού ε, παραβιάζοντα ε, το δίκαιο του ΠΟΕ, διακυβεύοντα την ασφάλεια. Έπειτα, η έκθεση αυτή θα πρέπει να καλωσορίσει την Συμφωνία Δευκόλυνση του Εμπορίου ω την πρώτη συμφωνία μετά τα τέλη τη δεκαετία του 90 που παρέχει αρκετή προστασία στο εμπόριο. Τέλος, ε, η συμφωνία για τις ε, δημόσιες προμήθειες ε, με την πολυμέρεια που τη διακρίνει θα είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς το άνοιγμα των αγορών αλλά και προς τον ανοιχτό διαφανή ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειες μαζί με τα μέλη του ΠΟΕ για να επιτύχει αυτή η συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπούχνερ εκ μέρου των Πρασίνων. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω λίγα σχόλια. Συμφωνούμε μεν ότι η έκθεση αυτή πρέπει να ε, παρουσιάσει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία. Όμως ε, θέλουμε να εμβαθύνουμε σε ορισμένα θέματα. Ε, να αναφέρω μόνο τον παράγραφο 5 για τα αίτια της παρούσας κρίσης. Παράγραφος 6 για μια νέα προσέγγιση που θα ε, διαφοροποιήσει την, ε, τα μέλη του ΠΟΕ που είναι εκβιομηχανισμένα και εκείνα που αναπτύσσονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί το σημείο αυτό. Διότι πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να ε, αλλάξουν προσέγγιση. Έπειτα, περισσότερο ευέλικτε διαπραγματεύσει πολυμέρεια στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ και με τη δυνατότητα συμμετοχή των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, κεφάλαιο 7, ενίσχυση του ΠΟΕ ως ενός οργανισμού που θα ε, αυξήσει την ε, διαφάνεια. Επίσης, παράγραφος 8 στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ε, προστασία του περιβάλλοντος και εδώ θέλει ορισμένες βελτιώσεις. Ελπίζουμε να ε, μας στηρίξετε για να πάμε τις ε, ιδέες και τη φιλοδοξία μας λίγο παραπέρα και εν της φωνίας με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ΓΚΟ, ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και τους δύο συγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει και για τους προβληματισμούς που εισήγαγαν σχετικά με την παρούσα κατάσταση του ΠΟΕ. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ είναι αναγκαία. Πράγματι χρειάζεται πολυμερής προσέγγιση. Έχουν δημιουργηθεί αρκετές ομάδες εργασίας ε, διεθνώς όμως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι το κέντρο της προσέγγισής μας. Χωρίς αυτές θα αποτύχει η διαδικασία πριν καν ξεκινήσει. Έπειτα, υπάρχει μία ευρεία συνένεση για την ατζέντα μετά την ανάπτυξη. Έγιναν οι σχετικές συζητήσεις και αυτό σημαίνει πως σε διεθνές επίπεδο υπάρχει ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και όταν συζητάμε για το θεματολόγιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να βλέπουμε λίγο πιο μακριά πώς δηλαδή θα πρέπει να λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία τον 21ο αιώνα. Εάν δεν συμπεριλάβουμε και αυτή την άποψη, της πολυμέρειας δηλαδή του εμπορίου, δεν θα ε, έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Σε 20-30 χρόνια θα έχουν αποτύχει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και με τους συζητητές έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι πτυχές αυτές, τρίτες πτυχές σε συνδυασμό με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ε, επίσης ε, συνδεδεμένα με την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Μιλτό Σαπάτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ήθελα να τονίσω ότι η συνολική κατάσταση με τον ΠΟΕ παραμένει δύσκολη. Όπως θα έχετε παρατηρήσει βρισκόμαστε σε προβληματική κατάσταση ε, με τα ελλειπή ε, εφαρμογή λόγω των αντιμετρών αλλά αυτό που συμβαίνει ότι όλο ένα και περισσότερο μεταξύ των μελών του ΠΟΕ συμφωνείται ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση και ότι πρέπει να προστατευτεί ΠΟΕ. ήταν καλή έκβαση της Υπουργικής. Ε, προέκυψε το συμπέρασμα ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί ο ΠΟΕ και εμείς φυσικά ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουμε το πολυμερές σύστημα και πρέπει να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή οποιασδήποτε μεταρρύθμισης και οποιασδήποτε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Θα είδατε το σημείωμα, ε, το ενημερωτικό της Κομισιόν το οποίο ήταν πολύ θετικά οι περισσότεροι εμπορικοί μας εταίροι. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ξεκινήσει να διαδίδουμε τις ιδέες που παρουσιάζουμε σε αυτό το έγγραφο στους εμπορικούς μας εταίρους. Σε ομόκεντρους κύκλους κατά κάποιο τρόπο. Πρώτα απ' όλα έχουμε την τριμηρή συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία, αυτό το μηχανισμό που πολλά από τα ζητήματα που έχουμε στο έγγραφό μας ε, έχουν τεθεί εκεί και έχουν ε, συζητηθεί και πολύ θετικά μάλιστα. Μετά έχουμε ε, κάποια άλλα σημαντικά μέλη μέσω των G20, ε, όπως ανέφερατε η Γερμανία. Ε, χτίζουμε κάποια πολιτική στήριξη με ευρύτερους κοινωνικούς εταίρους, ε, συγγνώμη, εμπορικούς εταίρους και μετά με τα μέλη στη Γενέβη. Θέλουμε μία διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε τα εμπόρια και κάποιες αμετακίνητες θέσεις που έχουν ε, μπλοκάρει άλλε περιπτώσει να μα μπλοκάρουν και τώρα. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασία ε, με την Κίνα στη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε η Κίνα να εμπλακεί στη διαδικασία αυτή. Επίση, έγιναν χρήσιμε συζητήσει με τα 12 μέλη του ΠΟΕ που συγκέντρωσε ο Καναδά σε επίπεδο υφυπουργών και αναμένουμε μια ωφέλιμη συζήτηση σε υπουργικό επίπεδο τον Οκτώβριο. Ωστόσο θα θέλαμε να εστιαστούμε όσον αφορά στις διάφορες προτάσεις, στη δική μας πρόταση, διότι η καναδική πρόταση είναι λιγότερο φιλόδοξη και λιγότερο εστιασμένη από τη δική μας. Για το σχέδιο έκθεσης ε, συμφωνούμε με τα βασικά μηνύματα και με τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για ενίσχυση του πολυμερού εμπορικού συστήματο και παραμένουμε και εμεί δεσμευμένοι για να προχωρήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ ω εισηγητή. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου για τα σχόλιά σα και αναμένω τι τροπολογίε σα, τη συμμετοχή σα. Ο συνεισηγητή μου. Κύριε Χάνσελ, θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν το σημείο αυτό. Προθεσμία τροπολογιών είναι η 11η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πάμε απευθείας στο σημείο 14. Πολύ σύντομο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Καρολίν Κράς Βάντερ Χάιντς είναι η συγκήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δώστε μου λίγο χρόνο σας παρακαλώ γιατί είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή πιστεύω και μεγάλη σημασία της. Αγαπητοί συναδελφοί, το τελευταίο διάστημα το εμπόριο δεν ταυτίζεται απλώς με την παγκοσμιοποίηση, αλλά μας ανησυχεί και πάρα πολύ. Ακόμα και αν οι ειδικοί και επιστήμονες, οι οικονομολόγοι λένε ότι γενικά είναι θετική η παγκοσμιοποίηση, ε, υπάρχουν ε, ορισμένοι κλάδοι που πλήττονται μειώνεται το εισόδημα, χάνονται θέσεις εργασίας, χάνονται τα κέρδη και δείχνει πραγματικότητα ότι πάντα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Και δεν κερδίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο σε μια κοινωνία ή σε περιφέρεια ή σε χώρα. Υπάρχουν ε, ανισότητες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές και στο παρελθόν ε, δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά, άρα εντάθηκαν ακόμα περισσότερο. Είναι κρίμα που στις εμπορικές συμφωνίες με την Ένωση, ε, της Ένωσης, ιδιαίτερα στα κεφάλαια ε, για την αηφορία. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να επιβάλλουν την προστασία ε, των ε, εργασιακών και των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Οι κυρώσει είναι η έσχατη καταφυγή, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση για να επιβληθούν και ελπίζω να έρθει αυτή. Ποιο είναι τώρα ο στόχο αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση να προστατεύονται οι εργαζόμενοι ε, άνδρες και γυναίκες που απολύονται λόγω της αυτοματοποίησης, της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Είναι πολύ μικρός ο προϋπολογισμός όμως και περίπλοκες οι διαδικασίες, αλλά παρόλα αυτά το συγκεκριμένο ταμείο για την παγκοσμιοποίηση έχει βοηθήσει πάνω από 140.000 απολυμμένους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι το Ταμείο αυτό δεν ε, εξαντλείται, δεν απορροφάται πλήρως. Τι προτείνω εγώ. θα πρέπει να μειωθούν οι διαδικασίες και να απλοποιηθούν για την υποβολή αίτησης και τα κράτη-μέλη ε, να υποστηρίζονται. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κόμβος όπου να ενημερώνει ε, τους ενδιαφερομένους. Ε, το άλλο θέμα είναι το πεδίο εφαρμογή. Θα πρέπει αυτό να ε, διευρυνθεί και να γίνει πιο ελαστικό, έτσι ώστε όσοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, αλλά και περιφέρειες που πλήττονται από τη συγκυρία από μια μεγάλη ε, ανεργία να μπορούν να ε, υποστηρίζονται. Και ένα άλλο σημαντικό, για τη βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης θα πρέπει να έχουμε καλύτερα ε, και περισσότερα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που συλλέγουν τα κράτη-μέλη. Το ποσοστό συγχρηματοδότηση θα πρέπει να αυξηθεί στο 70% για το ταμείο αυτό και είναι σημαντικό και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, ανεπτυγμένες δομές στην αγορά εργασίας τους να μην παραμελούνται και να συνυπολογίζονται, συμπεριλαμβάνονται. Ε, και στις εμπορικές συμφωνίες επαναλαμβάνω να υπάρχουν κεφάλαια με κυρώσεις για να ε, φτάσουμε στην φόρο ανάπτυξη, στις αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης και σωστές συνθήκες αγοράς. Το εμπόριο όμως δεν είναι διεθνές. Θα πρέπει τα έσοδα ε, αυτού του, του διεθνούς εμπορίου μάλλον να κατανέμονται καλύτερα και δικαιότερα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και ενδιαφερομένων και να παίζουν σημαντικό ρόλο και να έχουν λόγο η κοινωνία των πολιτών, η ΜΚΟΤΑ, συνδικάτα κτλ. για να υπάρχει καλύτερο συντονισμός και μεγαλύτερη συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά που ε, προτιθέμεθα να συνάψουμε εμπορική συμφωνία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύει εκ των προτέρων ε, τις συνέπειες ενδεχόμενες αυτής της συμφωνίας. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι σημαντικοί εταίροι ε, για τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να επωφελούνται όλοι. Και εκείνοι που δεν ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές υποχρεώσεις θα πρέπει να λογοδοτούν. Ξέρουμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία της αγοράς είναι βασικός πυλώνας του δικού μας οικονομικού μοντέλου και κοινωνικού μοντέλου και έχουμε σημαντικούς μηχανισμούς να αντισταθμίζουμε τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Περιμένω με χαρά τη συζήτηση και τις προτάσεις των συναδέλφων και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φουγούας από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει στο θέμα αυτό. Στόχο ήταν να διασφαλιστεί ότι το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να παρέχει ε, στήριξη οικονομική και αλληλεγγύη μετά το 2020 ο ανταγωνισμός ε, αυξάνεται, νέες προκλήσεις αναδύονται, γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεπεράσουμε τις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής και να εξετάσουμε πτυχές που ε, έχουν επίσης ε, σχέση με αυτό. Δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στα εμπορικά ζητήματα, σε εμπορικές πτυχές. Πρέπει να εστιάσουμε σε βασικούς τομείς. Βελτίωση της παρακολούθησης, ε, της χρήσης των κονδυλίων. Θέλουμε καλύτερα στοιχεία, θέλουμε αξιολόγηση αντικτύπου της χρήσης των κονδυλίων, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού, πρέπει να εξετάσουμε τις σχέσεις του με το ενδοενωσιακό εμπόριο διότι ενδεχομένως ε, ελοχεύουν αρτικές επιπτώσεις για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται ειδικές διατάξεις. Επίσης, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές ε, παγκόσμια στο εμπόριο, οι δομές που ενδεχομένως αλλάζουν και στηρίζουν το εμπόριο. Η καινοτομία της τεχνολογίας είναι επίσης πολύ σημαντική. Πρέπει να προσαρμόσουμε τους ε, κανόνες ε, με ή να δημιουργήσουμε καινούριου σύμφωνα με τις εξελίξεις και να φροντίσουμε να ε, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ε, νέες προκλήσεις. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα ήθελα να συμπεριληφθούν στην έκθεση και θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ με τους συναδέλφου έτσι ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Α, η Έμα. Παρακαλώ. Μιλώ εκ του κυρίου Λούνες. Η ομάδα στηρίζει απόλυτα τα μέτρα που έχουν τεθεί για τι ε, πολιτικέ που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσει απασχόληση. Ωστόσο, ε, πιστεύουμε ότι το Ταμείο Παρασαρμογή στην Κοσμοσπίση δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο, ούτε θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματικό ε, στην επανένταξη των απολυμένων εργαζόμενων στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται νέα, να ληφθούν υπόψη τα νέα κριτήρια, οι νέε τάσει ε, στο παγκόσμιο εμπόριο και να παρατηρήσουμε και να διορθώσουμε τις ασυμφωνίε με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ε, ιδιαίτερα εν ώψη μεγάλων αναδριαρθρώσεων. Αυτά έχουν να πούν η ομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ. Μια σύντομη παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον κύριο Λουσιάν Σεγνέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρου των υπηρεσιών τη Επιτροπή να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό το μέσο. Είναι ένα από τα πολλά που χρησιμοποιούμε για να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη σε διαφορέ περιοχές. Επιμένω στο ότι, όπως αποδείχθηκε στο παρελθόν, το Ταμείο αυτό έχει να παίξει σημαντικό ρόλο μεταξύ όλων των μέσων που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, Προφανώ τα δεδομένα είναι επαρκή και υποστηρίζω πράγματι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Είναι αναγκαίο να παρακολουθούμε πιο στενά και να βελτιώνουμε την εκ των υστέρων αξιολόγησή μα, την οποία ούτω ή άλλω έχουμε καταφέρει να κάνουμε και η οποία δείχνει αναμφίβολα ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή πολλών ανθρώπων που βρήκαν δουλειέ χάρη σε αυτό. Τα σχόλια φυσικά εστιάζονται στη βελτίωση, στην επέκταση του EGF, του Ευρωπαϊκού Ταμείου στην Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και στην καλύτερη προσαρμογή του στι πραγματικέ συνθήκε. Αλλά πολλά στοιχεία, κατά την άποψη τη Κομισιόν, δεν έχουν εξισορροπηθεί πολύ σωστά στην παρουσία του μορφή. Για παράδειγμα, η ικανότητα του Ταμείου να παρέχει απευθεία κονδυλία στι ε, περιφέρειες. Αυτό δεν συνάδει με το πνεύμα του Ταμείου, διότι το Ταμείο αυτό ε, από σκοπή στο να βοηθά εργαζομένους, όχι περιφέρειες. Έχουμε άλλα μέσα που μπορούν να διοχετεύσουν κονδύλια σε περιφερειακές αρχές και σε περιφέρειες. Ε, φυσικά, αν οι περιφέρειες θέλουν να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία, αυτό μπορούμε να το δούμε. Αλλά τα χρήματα αυτά υποτίθεται ότι προορίζονται για τη βοήθεια επιμέρους εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους. Ε, Επίσης υπάρχει κάποιο πρόβλημα συνοχής μεταξύ κάποιων τροπολογιών και των μέτρων και των εξάντε και του εξπόστ. Το ταμείο αυτό έχει σχεδιαστεί ως ταμείο εκ των υστέρων, όχι εκ των προτέρων. Δηλαδή δεν λειτουργεί προληπτικά, προορατικά. Λειτουργεί αφού δημιουργηθεί το πρόβλημα. Γιατί προβλέψεις, δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε ποιο θα χάσει τη δουλειά του σε ποια περιοχή και πόσα, για πόσα χρόνια και να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα το Ταμείο. Δυστυχώ, οι προτάσει αυτέ που κάνετε σχετικά με αυτό δεν είναι εφικτέ. Ευχαριστώ. Άρα φυσικά ξέρετε το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν αυτό δυσαρεστεί την Κομισιόν. Ε, παραδοσιακά έτσι κάνουμε εδώ και χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ λόγω του ότι η γνωμοδότηση ε, αυτή απευθύνεται στην ε, ε, πρέπει να βιαστούμε διότι έτσι είναι η διαδικασία δηλαδή σήμερα 27 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα μπορείτε, είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών θέλετε να πείτε κάτι Καρολίν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξο βέβαια το χρονοδιάγραμμα για αυτό το σημαντικό θέμα. Σύντομα μόνο να πω ε, κάτι για τις περιφέρειες. Είναι σημαντικό να διευρεθεί το πεδίο εφαρμογής και αν συμμετέχουν και τα συνδικάτα και άλλοι ενδιαφερόμενοι στην προσπάθεια αυτή, είναι και προ όφελο των απολυμένων. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνω πρόταση, γιατί έχουν πρόβλημα οι μικρομεσαίες να αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση και τις ανετικές της συνέπειες. Το ταμείο αυτό δεν ε, εξαντλείται στην απορρόφηση, άρα χωράει βελτίωση και ευελιξία για να μπορούν ε, να υποφελούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Εξού και προτείνουμε το συγκεκριμένο κόμβο, αυτό το hub desk. Κρίμα που είναι το μόνο που έχουμε, αλλά βελτιώσει χωράει πάντω. Ευχαριστώ για την καλή συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία λοιπόν σήμερα το απόγευμα στι 6 μόνο στα αγγλικά τροπολογίε, έτσι έχουν συμφωνήσει οι πολιτικέ ομάδε. Τελευταίο σημείο 15 παρουσίαση του εγγράφου θέσης του εμπορικού επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα. Καλωσορίζω τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, Ματς Χάρμπορν, και θα του δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε και ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω πέντε λεπτά για την παρουσίασή Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τον έγγραφο θέση. Πολύ σύντομα, είναι ένα από τα τρία έγγραφα παρουσιάσαμε φέτος. Ε, παρουσιάσαμε μία έρευνα ε, σε ένα συνέδριο και τι έγινε στους 18 μήνες μετά ε, την μεταρρύθμιση που μας υποσχέθηκαν. Σημειώσαμε αυτά που έγιναν τους τελευταίους 18 μήνες. Δεν περιμέναμε και πολλά, είναι η αλήθεια, ε, από την Κίνα. Μετά τις πολιτικές όμως συναντήσεις που είχαμε την Κίνα, είδαμε κάποια πρόοδο και είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ακριβώ, διότι η πρόοδο συντελείται επειδή η Κίνα το επιθυμεί, αλλά και επειδή τα θεσμικά όργανα και το επιμελητήριο ε, εργάστηκαν σκληρά. Βέβαια, δεν θα σα μιλήσω για την πρόοδο, αλλά θα εστιάσω στα προβληματικά σημεία. Πρώτο προβληματικό σημείο είναι και ένα σημείο που είδαμε πρόοδο. Πρόσβαση στην αγορά. Όπως θα παρατηρήσατε όλοι, η Κίνα αυτή τη στιγμή άρει τους περιορισμούς σε πολλούς τομείς, σε χρηματοοικονομικά, ασφάλειες, ναυπηγεία. Ναι, κοινοπραξίες Επίσης, η Κίνα έχει μειώσει τον αρνητικό κατάλογο και τώρα είναι 48 απαγορευμένοι περιορισμένοι τομεί. Ε, μας ανησυχεί βέβαια ότι αυτός ο στόχος δεν είναι αρκετά φιλόδοξος, ότι οι διαπραγματεύσεις ε, πρέπει να συνεχιστούν για μια ολοκληρωμένη συμφωνία επενδύσεων. Βέβαια, Ακόμα δεν έχουμε δει τι μα προσφέρει η Κίνα σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά. Χρειάζεται όμω περισσότερη φιλοδοξία έτσι ώστε να συντελεστεί πρόοδο. Τώρα, σε σχέση με τα ανοίγματα πρόσβαση στην αγορά, τι μας κρατάει πίσω. Η υπερβολική ρύθμιση που δεν ε, διευκολύνει, που εμποδίζει την πρόσβαση. Από την πλευρά της Κίνας επίσης ένα πρόβλημα είναι το θέμα της χορήγησης αδειών ε, στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ακόμα είμαστε εξαρτημένοι από τη χορήγηση αδειών και αυτές δεν χορηγούνται εύκολα. Πώς συνεχίζουμε. Το πιο σημαντικό θεωρούμε πως είναι να συνεχίσουμε το διάλογο με την Κίνα. Μόνο έτσι θα μεταρρυθμιστεί το ε, ρυθμιστικό, υπερβολικά ρυθμιστικό περιβάλλον της Κίνας. Και θα έχουν νόημα οι προσπαθίες μας. Τώρα, αν συγκρίνουμε τα δύο αυτά ζητήματα, πρόσβαση στην αγορά και ρυθμιστικές ετάσεις με την Ευρώπη, ε, θα σταθούμε στον τομέα της κυβερνασφάλειας και της τεχνολογίας πληροφορικής ε, και επικοινωνίας. Πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά επηρεάζεται και ε, η μελλοντική ψηφιακή ε, μετάβαση. Χρειάζεται λοιπόν δημιουργία νέα στρατηγική μαζί με την Κίνα το συντομότερο. Για περισσότερη πρόσβαση στην αγορά από εταιρείε, περισσότερη πρόσβαση σε τεχνικές επιτροπές και σε ε, διάφορα φόρα όπου ε, συζητούνται οι τεχνικές αυτές αλλαγές. Είναι ένας τομέα στον οποίο πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε. Άλλη προβληματική τομείς, από ό,τι φάνηκε από το συνέδριο, είναι η συνέχιση των διακρίσεων ε, εις βάρος των ξένων επιχειρήσεων στην Κίνα. Αυτό δεν είναι πάντα κρατική πολιτική, αλλά και προστατευτισμό σε τοπικό επίπεδο. Τα κύρια αίτια αυτών των διακρίσεων είναι ο ίδιος ορισμός μιας εταιρείας ε, ξένων επενδύσεων. Εμείς έχουμε προτείνει η Κίνα να καταργήσει τον ε, νόμο αυτό, το οποίο θα εξαφάνισε και αυτήν την διάκριση που δημιουργεί προβλήματα. Μετά, κρατικές επιχειρήσεις στην οικονομία της Κίνας. Στο πολύ καλό έγγραφο σχετικά με τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, παρατηρούμε ότι ναι, μεν γίνονται μεταρρυθμίσεις στη χώρα, όμως με πολύ περισσότερη διαφάνεια από την αναμενόμενη, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαστρεβλώσεις στην οικονομία εξαιτίας αυτού. Επίσης, ζητούνται σαφή χρονοδιαγράμματα. Όλα αυτά για μας συνιστούν το έλλειμμα μεταρρυθμίσεων. Βλέπουμε ότι η Κίνα μεν οριμάζει, μεγαλώνει, προχωρά, δεν προφταίνει όμως την ορίμανση ε, της συγκυρίας. Μόνο μέσω των μεταρρυθμίσεων θα αμβλημθούν οι εντάσεις που παρατηρούνται παγκόσμια. Τώρα να επανέλθω στο έγγραφο, εξαιρετικό έγγραφο, σημείο 1 πολύ σημαντικό να υπάρχουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν ευκαιρίες για επικοδομητικό διάλογο. Θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αρκετοί πόροι έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά όργανα να μπορέσουν να εισέλθουν σε έναν επικοδομητικό διάλογο με την Κίνα. Και ως ε, εταίρος έχουμε και ευθύνη ιεράρχησης των προτεραιοτήτων έτσι ώστε να δαπανίσουμε πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος, η πρωτοβουλία Μία ζώνη, ένας δρόμος. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ενωμένη στρατηγική απέναντι στην Κίνα. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε την πρωτοβουλία έτσι ώστε αυτή να γίνει περισσότερο διάφανη και να ε, ιδιαίτερα στον τομέα των ε, δημόσιων ε, διαγωνισμών. Τώρα, η εμπορική διαμάχη Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Τι συμβαίνει εδώ. Πράγματι, στην έρευνά μας είδαμε ότι πάνω από το 90% των ε, συμμετέχοντων χωρών ήταν αναγκασμένες να εκφράσουν ανησυχίες. Ωστόσο, το έγγραφο 19, το οποίο απαγορεύει οποιαδήποτε επίσημη ε, Οπότε επίσημη μεταφορά τεχνολογίας προς την Κίνα δείχνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα κακοδιαχείρισης από τεχνολογικές εταιρείες ε, με την εξαναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση της Κίνας εννοεί τις ε, μεταρρυθμίσεις που θέλει να κάνει είναι ειλικρινή ω προς τις προθέσεις της και εμεί θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται ε, όταν προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες των μεταρρυθμίσεων. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Σας ευχαριστώ και εγώ και τώρα θα δώσω το λόγο ε, στο συντάκτη αυτής της εξαιρετικής έκθεσης, ε, τον κύριο Βίνκλερ, το μόνιμο εισηγητή μας. Πραγματικά, εμείς είμαστε πολύ ισχυρή επιτροπή. Μπορούμε να λύσουμε το συνικό πρόβλημα σε 15 λεπτά. Κοιτάξτε πόσο φοβερή και τρομερή επιτροπή είμαστε. Οι ε, σχέσεις μας εμπορικές και οικονομικές είναι όλο και περισσότερο θέμα ισορροπίας. Content to, to give to our uh, international... Λοιπόν, ε οι ευρωπαϊκές, ευρωσυνικές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και επίσης ε, όλο και περισσότερο γιατί ε, είμαστε ε, ενός, μάλλον στα μέσα ενό εμπορικού πολέμου, ούτε καν στην αρχή, σοβεί ο πόλεμος. Έχει γίνει πρόοδος ε, βέβαια από τους Κινέζους φίλους μας, θα πρέπει να τον αξιολογούμε ε, σωστά, αλλά και ταυτόχρονα λέμε και ποια θέματα μας ανησυχούν. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Χάρμπορν, και το ανέφερα σημαντικότερο θέμα ανησυχίας, ε, το κείμενο ασφάλεια και οι τεχνολογίες τεχνολογι... Ε, επικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό αφορά τις παγκόσμιες σχέσεις, τις οικονομικές και το εμπόριο, όχι μόνο τις ευρωσυνικές. Ε, έχουμε αρκετά θέματα που μας ανησυχούν, οι ίσοι κανόνες παιχνιδιού, η ίση μεταχείριση των ξένων επενδυτών και των τόπιων επιχειρηματιών, θέματα πνευματικής πνευματικής ε, ε, ιδιοκτησίας, αναγκαστικής μεταφοράς, τεχνολογίας κτλ. Ε, είναι σημαντικό να ακούσουμε το επιμελητήριο αυτό στην Επιτροπή μας, γιατί έχει πολύτιμη εμπειρία για μας. Ε, το είδαμε αυτό και στην αντιπροσωπεία μας όταν είχαμε μεταβεί στην Κίνα. Ήταν πάρα πολύ κρίσιμο το επιμελητήριο για να καταλάβουμε τις νέες πραγματικότητες στην Κίνα. Να συνεχίσουμε φυσικό να εργαζόμαστε με την Κίνα, να συνεργαζόμαστε για αυτά τα θέματα και για πολλά άλλα. Και αν κοιτάξουμε λίγο πίσω, ε, τι μας δείχνει η εμπειρία μας, ότι δεν έχει νόημα να ε, κατηγορούμε την Κίνα ε, και να ε, την δεν έχουμε απέναντί μας και να συγκρούμαστε. Αυτό δεν βοηθάει. Ίσα ίσα τη στρέφει στον αντίθετο δρόμο και δεν είναι καθόλου τα δικά μας συμφέροντα αυτά. Ένα λεπτό, κύριο Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ για την ενημέρωση, αλλά έχω δύο ερωτήσεις πώς έχει αυτή τη στιγμή η συνεργασία μας στην τεχνητή νοημοσύνη και στις νέες τεχνολογίες. Πού βρίσκεται και ποια είναι η κεντρική ιδέα και ο πυρήνας. Και δεύτερον, πώς επηρεάζουν οι αμερικανοσυνικές σχέσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Κίνα. Υπάρχει άμεσος αντίκτυπος. Ένα λεπτό και η απάντηση. Χαιρόμαστε που ε, βλέπουμε ότι ε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας ε, στην Ευρώπη για να καλύψουμε το κενό που έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα. Θα πρέπει να ζητήσουμε πρόσβαση να έχουμε και σε περισσότερες ομάδες εργασίας για να συζητούμε ευρύτερα ζητήματα και ζητήματα δεοντολογίας με τους Κινέζους φίλους μας. η σύγκρουση ε, Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας, μπορεί βραχυπρόθεσμα να ευνοήσει τις δικές μας επιχειρήσεις, αν και εμείς δεν θέλουμε έτσι να συναλλασσόμαστε. Θέλουμε η Κίνα να γίνει ένα χώρος ε, εμπορίου με ίσους κανόνες, ίδιους κανόνες για όλους. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες τώρα. Ορισμένες εταιρείε ε, κάποιων κρατών μελών χρειάστηκε να μετεγκατασταθούν και άλλες να ε, δουν ε, τι θα γίνει με τις, ε, τα παραρτήματα που έχουν εκεί. Εμείς θέλουμε να έχουμε επικοδομητικό διάλογο και όχι συγκρούσεις. μάλιστα. Και αυτό θα μπορούσε να είναι και γνώμονας για τη μελλοντική μας εργασία. Συνεργασία και όχι σύγκρουση. Εδώ ολοκληρώνεται και το σημείο 15. 16 είναι διάφορα, έχουμε κανένα διάφορο, όχι. Επόμενη συνεδρίαση 10 και 11 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σκληρή δουλειά που κάνετε εδώ στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και χαίρετε.